Συνάδελφοι, παρακαλώ. Σα είδα και στην κοινή συνεδρίαση Econ Badge, αλλά θα σας ευχηθώ καλή χρονιά και στη δική μας συνεδρίαση, που είναι η τακτική της δικής μας Επιτροπής. Καλώς ήρθατε. Ένα σας παρακαλέσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Πρακτικά των συνεδριάσεων της 9ης Νοεμβρίου 2016 και 28-29, 5 Δεκεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου. Ωραία. Κάποιες ανακοινώσεις. Να θυμίσω στα μέλη ότι μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα λάβει χώρα στο 3C050 αμέσως μετά τη δική μας συνεδρίαση σήμερα το πρωί και κατά την κοινή συνεδρίαση οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την πρόληψη του χρηματοοικονομικού συστήματος για σκοπούς λεύκανσης προσόδων για χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων θα ε, εξεταστούν εκεί. Επίσης ε, για τους τριμερείς διαλόγους, πρώτος γύρος 15 Δεκεμβρίου. Το Κοινοβούλιο παρουσίασε τις τροπολογίες του περαιτέρω. Φαίνεται να υπάρχει προθυμία για να συμπεριλάβουμε στοιχεία για την ε, βελτίωση της ε, διατύπωσης. Αλλά η θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ιδίως για την ΕΙΟΠΑ και το EFRC είναι θέματα που δεν επιλύθηκαν, οπότε η Προεδρία θα δει τι μπορεί να γίνει από τα κράτα μέλη μέχρι τον επόμενο τριμερή διάλογο. Και ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό στα τέλη Μαρτίου 2017. Κάποιες αποφάσεις ε, από τη συνάντηση των συντονιστών το Δεκέμβριο κανονισμό για την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης ε, στο επίπεδο του Υπηρεσία για το ΦΠΑ, οδηγία για τι ε, εντατικότερε φορολογικέ υποχρεώσει. οδηγία για τα ποσοστά ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικών, PPP, οδηγία για εξαίρεση αντιστροφής του ΦΠΑ για ορισμένα κράτη-μέλη CCP, που απαιτεί ε, την σύμφωνη γνώμη των σοσιαλιστών και συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ε, έκθεση ιδίας γνώμη πρωτοβουλίας των ε, σοσιαλιστών. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε στην Επιτροπή Εικόνη για τον τοσχέ της αφαρικιότητας που καθήλυνα αρμόδια <clears throat> είναι άλλη επιτροπή και μετά και οι συστάσεις για τις αναχώρα ε, η αναχώρα μάλλον συστάσεις. Εδώ δεν έχουμε άλλα νέα. Μάλλον υπάρχει και οικονομική διακυβέρνηση. Συμφωνήθηκε ο κύριος Ντάισεμπλουμ να έρθει στην Επιτροπή Οικονομικών νωρίτερα από ό,τι είχε προτείνει το γραφείο των συνεργατών του. Ζητήθηκε ε, έκτακτη συνεδρίαση λοιπόν και ο Διευθυντής της Ταλική Κεντρική Τράπεζα θα έρθει σε μια έκτακτη συνεδρίαση για το 2017 η Επιτροπή θα έρθει στην ΕΚΟΝ την ίδια μέρα ή την επομένη μετά τη δημοσίευση του σχεδίου προπολογισμού. Οι συντονιστοί θεώρησαν ότι το χρονοδιάγραμμα την προηγούμενη χρονιά ήταν πολύ αργά και θα έρθουμε σε επαφή και με τη Γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού για να δούμε μαζί με τους Ευρωπαίους ε, υπευθύνου ε, του SSM και ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης θα προσκληθεί για να δούμε την υλοποίηση της έκθεσης Γκουλάρ για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού για του χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Ευρώπη. Αυτέ οι ανακοινώσει. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Εξέταση τροπολογιών τη έκθεση του κ. Χόκμαρκ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κύριε Σιγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ σε όλου καλή χρονιά. Με όσα συμβαίνουν στον κόσμο μα, θα το χρειαστούμε. Ε, η έκθεση αυτή έχει λάβει 500 περίπου τροπολογίε, 593 για την, 593 για την ακρίβεια. Πάρα πολλέ. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει πολλέ φορέ για τα ίδια άρθρα. Δηλαδή κάποιε φορέ φαίνονται περισσότερε τροπολογίε από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Αλλά είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον των συναδέλφων και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστούμε με του ε, σκιώδει. Είχαμε κάποιες πρώτες συζητήσει και να πω τη από τη δική μας πλευρά η εξέταση όλων αυτών των τροπολογιών σε αυτούς τους καιρούς αβεβαιότητας που περνάμε Βλέπουμε τι συμβαίνει στι ΗΠΑ, βλέπουμε τι συζητήσει για το Brexit και τι ακούμε. Τη χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική αστάθεια από όλα τα κράτη-μέλη μα, πολλέ από τι προκλήσει και τα προβλήματα που μα ταλανίζουν. Νομίζω ότι το σύμφωνο σταθερότητα είναι ε, ακόμη πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση, διότι δίνει αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και αν υπάρχει ω προ αυτό έλλειψη εμπιστοσύνη, μπορεί να υπονομευτεί η ίδια μα η σταθερότητα. Μια ζωτική σημασία σε ερώτηση για τι διαπραγματεύσει που θα έχουμε είναι πώ να εκλάβουμε αυτό που έχει ονομαστεί θετική δημοσιονομική στάση Είμαι πάντοτε θετικός ω προ τα θετικά πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, εάν μπορούμε τα ε, κρατικά δημοσιονομικά να τα προστατεύσουμε, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη, είναι σημαντικό αυτό. Είναι καθήκον μας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα είδος συμφωνίας όλοι μαζί, με σεβασμό για το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά χωρίς να αφήσουμε δικαιολογίε για να υπονομευθεί η δημοσιονομική μας σταθερότητα. Και ταυτόχρονα να βεβαιωθούμε ότι τα δημοσιονομικά κίνητρα που διατίθεται μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε σε ένα πλαίσιο ευελιξίας, αλλά μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας. Και να επιτρέψουμε να δοθούν και ευκαιρίες για ποσοτικοποίηση το σχεδιασμό του προπολογισμού. Πρόεδρε, πάντοτε με εκπλήσει όταν οι συζητήσει για σημαντικέ δαπάνε φέρνουν του συναδέλφου τη κυβέρνηση να λένε ότι αυτέ οι δαπάνε είναι πιο σημαντικέ από κάτι άλλο. Γι' αυτό πρέπει να υπερβούμε τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητα. Μα είναι τόσο σημαντικέ αυτέ οι δαπάνε, πρέπει κανεί να ξεκινήσει από αυτό πριν ξεπεράσει τα όρια Δηλαδή να είναι η πρώτη δαπάνη που θα προβλεφθεί. Όχι στο τέλο του σχεδίου των προπολογισμών να ε, προστίθεται και να πούμε ότι πρέπει να υπερβούμε τα όρια. Όχι. Νομίζω ότι αυτό ο τρόπο κατηγοριοποίηση των δαπανών θα μα επιτρέψει να πετύχουμε πολλά καλά αποτελέσματα. Αυτή θα πρέπει να είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Και είναι και αυταπόδεικτο. Διότι έχουμε τη σχετική νομοθεσία την ε, εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι και καθήκον τη να επιβλέπει ότι εφαρμόζεται αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε πολύ. Και ε, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία και να συνεννοηθούμε για το πώ όλα αυτά μπορούν να επιδιωχθούν. Ε, πρέπει να δούμε πόσε πολλέ τροπολογίε ασχολούνται με το θέμα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Τα πράγματα διαφέρουν από κράτο μέλο σε κράτο μέλο προφανώ. Πολλοί συνάδελφοι επισημαίνουν ότι υπάρχει ανισότητα ή άνηση κατανομή τη οικονομική ανάπτυξη ή τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Εγώ δεν θεωρώ ότι γίνεται βάσει σχεδίου αυτό. Προκύπτουν και προχωρούμε. Ε, είναι διαφορετικέ οι περιστάσει κάθε φορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Έχουμε κάποια ανάπτυξη σε κάποια κατημέλη. Μεγαλύτερη σε κάποια, μικρότερη σε άλλα. Και αυτό έχει να κάνει και με τις πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα. Νομίζω αυτό πρέπει να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε. Πρέπει να δούμε τα συνολικά στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη μια, αλλά από την άλλη και τις επιμέρους ε, καταστάσεις και τα επιτέγματα του κάθε κράτους μέλους. Πρόεδρε, αν βάλει κανείς το κεφάλι του στο ψυγείο και τα πόδια του στο φούρνο, Προφανώς θα είναι διαφορετική η θερμοκρασία του. Και ο μέσος όρος θα είναι καλός. Αλλά αυτό δεν είναι καλό ούτε για τα πόδια του για το κεφάλι ταυτόχρονα. Και αυτό είναι σημαντικό και στις οικονομικές πολιτικές. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε το σωστό. Και ότι έχουμε ανάπτυξη και θέσει εργασία μεν. Ο συντονιστής βλέπω αντιδρά. Αλλά Σίγουρα οι διαφορετικέ περιστάσει ε, οδηγούν σε διαφορετικέ ευκαιρίε. Οι επενδύσει για μα είναι πολύ σημαντικέ. Και οι επενδύσει γενικώ προσελκύουν και άλλε επενδύσει. Δημιουργούν ένα αίσθηση ότι υπάρχει δυνατότητα κέρδου, που είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό επίση ότι από διαφορετικέ ομάδε πολλά μέλη τονίζουν την ανάγκη για χαμηλότερου φόρου και περισσότερε θέσει εργασία. Καλό αυτό. Όταν συζητάμε τι διαδοτικές μεταρρυθμίσει επίση. να ολοκληρώσω εδώ τη σκέψη μου. Αυτό προκύπτει και από τις περισσότερες τροπολογίες. Τι έχουμε εδώ, χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη, βραδίτητα δηλαδή, που έχει να κάνει με τα έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής των τελευταίων ετών. Αυτό δεν είναι βιώσιμο όταν θα υπάρξει μια σταδιακή μείωση αυτών των μέτρων, θα πρέπει να βασιστούμε στι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Βεβαίω, μπορούμε πάντα να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν δημοσιονομικά κίνητρα. Όμω, ε, αυτό το περιμένουμε στι ευρωπαϊκέ οικονομίε εδώ και πολύ καιρό. Και ό,τι άποψη και να έχουμε, δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε ήδη δώσει υπερβολικά πολλά δημοσιονομικά κίνητρα. Εδώ πρέπει να υπάρξουν λοιπόν διαφορετικέ μεταρρυθμίσει και υπό αυτή την προοπτική. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, διότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τα κρατικά δημοσιονομικά, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προσελκύσουν επενδύσεις, πρέπει να έχουμε σταθερότητα και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα τρία στοιχεία, αυτές οι τρεις παράμετροι μπορούν να συνδυαστούν. Η θετική δημοσιονομική στάση ε, θα μα βρει ευνοϊκά διακείμενο εφόσον είμαστε θετικοί στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Λέει ο πρόεδρο Κουαρτιέρη, ο κ. Σίλβα Περέιρα, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ να ευχηθώ σε όλου του συναδέλφου καλή χρονιά να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Μάρκε για την ε, παρέμβασή του, την παρουσίασή του και να δηλώσω την προθυμία των σοσιαλιστών να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να καταλήξουμε σε μια συναντητική πρόταση. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Η τωρινή εκδοχή της έκθεσης απέχει αρκετά από το σημείο που θα μας επέτρεπε να καταλήξουμε σε συνένεση. Δεν υπάρχει όμως λόγος να αμφιβάλλουμε ότι το πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας που μας διέπει θα μας επιτρέψει, όπως και στο παρελθόν, να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση. Ως εκ τούτου. Οι ε, συμβαστικέ λύσει που έχουν βρεθεί σε προηγούμενε περιστάσει θα πρέπει να είναι ένα σημείο αναφορά. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση είναι σε αυτή τη φάση το Ευρωκοινοβούλιο να μειώσει τις φιλοδοξίες του σε σχέση με το παρελθόν, ιδίω ως προς τις προϋποθέσεις για την δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη στον χώρο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εκδηλώνω επισήμω τη διάθεσή μου να συνεργαστούμε, αλλά και να αναφερθούμε σε προσπάθειες και εκθέσεις που έχουν ε, προκύψει τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα μας θέλει να συζητηθεί το πρόβλημα τη αξιοπιστίας των κανόνων ή τουλάχιστον να έχουμε κανόνες αξιόπιστους στη λειτουργία της Οικονομικής και Ένωσης. πρέπει να δούμε με προσοχή τα προβλήματα της Ευρώπης και ίσως το πρώτο που θα πρέπει να αναφέρουμε δεν είναι η αξιοπιστία των κανόνων ακριβώς. Το σοβαρό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έλλειψη επενδύσεων, η έλλειψη ανάπτυξης, η ανεργία, οι ανισότητες και οι διαφορές, οι ανισότητες. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και επειδή προκαλούν δυσαρέσκεια και κίνημα ε, διάλυσης ε, και εξάρθρωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, αυτή τη στιγμή ακριβώς βλέπουμε να τίθεται να αμφιβόλο η ίδια επιβίωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αυτό πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και να δράσουμε. Εδώ θα συμφωνήσω με τον εισηγητή όταν λέει ότι το αντικείμενο εδώ είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κάνουμε το σωστό η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι ορθή. Αυτή είναι αποφασιστική, γι' αυτό είναι αποφασιστική η στιγμή που ζούμε, συνάδελφοι. Είναι στη, αποφασιστική ω προ την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι αυτή η στιγμή όπου το, το, όπου το Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί ω προ την κατεύθυνση τη ε, οικονομική πολιτική και τη δημοσιονομική. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ένα ουσιαστικό πολιτικό γεγονός στο οποίο θα πρέπει να θεμελιώσουμε τη συζήτησή μα. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει στα κατημέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι το εξή. Η ευρωπαϊκή οικονομία ήδη από το 2017 θα χρειαζόταν μια δημοσιονομική πολιτική που να συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αυτό είναι η ανάγκη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δημοσιονομική πολιτική που να ε, συμπληρώνει και να συμβαδίζει με την νομισματική πολιτική. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή δεν μπορεί να παραμείνει εσαή με αυτή την εκτατική ορμή που είχε τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια λέει και κάτι ακόμα λέει ότι οι προπολογισμοί για το 2017 που μόλις ενέκρινε η υλοποίηση των ίδιων των δικών της, των συστάσεων για την επόμενη χρονιά θα οδηγούσαν σε δημοσιονομική πολιτική που θα είναι σχετικά περιοριστική και σχετικά εκτατική. Αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρώπη το 2017 θα ακολουθήσει σφαλμένη δημοσιονομική πολιτική, εάν δεν κάνουμε κάτι εδώ μεταξύ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση, αυτή που έχει γίνει γνωστή ως positive fiscal stance, θετική δημοσιονομική στάση, μια προσέγγιση πιο θετική δηλαδή, ώστε τα κράτη με περισσότερο περιθώριο στον προπολογισμό τους να κάνουν περισσότερα και για την ανάπτυξη. Πρόεδρε, συνάδελφοι, πιστεύω ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να αποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και να χαιρετήσει αυτή την πρόταση στηρίζοντάς την. Η δουλειά της ομάδας μας θα πρέπει να λάβει την κατεύθυνση της στήριξης όλων των μηνυμάτων που σκοπό έχουν να δώσουν έμφαση στην σημασία των επενδύσεων, ε, να καταπολεμήσουν τις ανισότητες και αποκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέψουν να σχεδιαστεί μια δημοσιονομική πολιτική που να βρίσκεται στο ύψος των προκλήσεων αυτής της ε, φάσης, της χρονικής περίοδου. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία αντίφαση με προηγούμενε τοποθετήσει και κινήσει του Κοινοβουλίου ή επιβολή κυρώσεων λόγω χάρη, δεδομένου ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε τέτοιε περιπτώσει. Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο, την κατάλληλη πολιτική ανάμειξη μέτρων, ε, το policy mix που θα επιτρέψουν να έχει μια καλή συνεισφορά και η δική μα ομάδα και όλη η Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματο του Ρόμπερτ Ζήλε, συναδέλφου μου, ο οποίος δυστυχώ κολλείεται σήμερα. Έτσι λοιπόν λέει ο κύριο Ζήλε. Έχουν κατατεθεί πολλέ τροπολογίε για την έκθεση ίδια πρωτοβουλία του κ. Χέκμαρκ που βάζει μια καλή κατεύθυνση αλλά χρειάζεται ακόμα κάποιες διορθώσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Με τις τροπολογίες μας θέλουμε να τονίσουμε ότι παρόλο που έχει επανέλθει η ανάπτυξη, είναι πολύ έφραστη και αργή και μεγάλες αποκλήσεις ανάμεσα στις χώρες μέλη. Το για την απασχόληση. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην απασχόληση μεταξύ των χωρών μελών. Πάντως, συνολικά μέτρα για την Ευρωζώνη ίσως κρύψουν κάποιες πραγματικότητες. Και υπάρχουν, όπως είπα, μεγάλες αποκλήσεις και στα ελλείμματα και στα χρέη κτλ. Ε, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι τα επίπεδα επενδύσεων. Αφενός μιλούμε για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Έχουμε και το σχέδιο Γιούνκερ που πολλοί θεωρούν πανάκια για την επίλυση όλων των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από τα χρήματα αυτού του σχεδίου όμως έχουν πάει σε χώρες που είχαν ήδη επαρκή επίπεδο επενδύσεων. Ενώ 13 ε, από τις χώρες Ευρωζώνης έχουν μόνο το 30%. Χρειάζεται να γίνουν και άλλες ε, τροποποίησεις. Εκφράζει τέλος την επιθυμία ο συνάδελφός μου να συνεργαστεί στενά με τον ε, εισηγητή και με του άλλους, άλλους σκιώδεις εισηγητές. Ε, βέβαια μόνο δύο λεπτά πήρα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω λίγα προσωπικά σχόλια. Ιδίω με την παρατήρηση ότι πολλά από τα χρήματα του EFSI κατευθύνθηκαν σε χώρες που είχαν ήδη επαρκές επίπεδο επενδύσεων. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις εξαρτώνται από το περιφερειακό προϊόν του κεφαλαίου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν αυξάνεται αυξάνοντας το κεφάλαιο, δηλαδή την προσφορά κεφαλαίου. Αντίθετα μάλιστα, για να αυξηθεί το περιφερειακό προϊόν του κεφαλαίου πρέπει να ενισχυθούν οι συμπληρωματικοί παράγοντες της παραγωγής το ανθρώπινο κεφάλαιο, η πρόσβαση στην τεχνολογία, η ποιότητα των υποδομών, η ποιότητα των δημόσιων διοικήσεων. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν το προϊόν του κεφαλαίου. Και εκεί υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες μέσα στην Ένωση, αφενός ανάμεσα στην παραγωγικότητα αυτών των συμπληρωματικών παραγόντων και των τιμών τους και την παραγωγικότητα σε σχέση με τις τιμές αυτές στις ε, του κέντρου της Ευρωζώνης και στις περιφερειακές από την άλλη μεριά. Επομένως, οδηγούμεθα σε διαφορετική κατανομή επενδύσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης. Άρα, το ζήτημα είναι ανταγωνιστικότητα. Επενδύσεις δεν πάνε σε χώρες που δεν είναι ανταγωνιστικές. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Ένα κρίσιμο πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν έχουμε πλέον τις ε, συναρματικές ισοτιμίες οι οποίες εξισορροπούν την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Επανερχόμεθα λοιπόν στο ότι το ευρώ είναι ακατάλληλο νόμισμα για μια ευρωπαϊκή ζώνη. Αυτά, ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ. Βιαντίχ από τους ελευθέρους. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι ευτυχισμένο 2017. 17. Ευχαριστώ κύριε Χακμάρκ για την έκθεσή σας, την οποία υποστηρίζουμε. Έχουμε υποβάλει ορισμένε τροπολογίες που είναι σημαντικέ για μας, για τις επενδύσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει τις προσπάθειες για να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα, εφαρμόζοντας και ενισχύοντας single market regulation όπως για τις κεφαλαιαγορές. Εμείς περιλαμβάνουμε στις τροπολογίες μας και συγκεκριμένες συστάσεις. Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για ε, τις επιχειρήσεις, οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της παιδείας, των ε, τεχνολογιών κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να προσελκύσει χρηματοδότηση για διαμεθοριακά ε, έργα σε όλη την Ένωση, για παράδειγμα μέσω του EFSI. Τώρα για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν συστάσεις αναχώρα χώρα και πρέπει να ολοποιούν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση ενιαίας αγοράς. Αυτά εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες για την φροντίδα υγείας. Για παράδειγμα με την ε, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δαπάνε υγεία στι χώρε μέλη είναι μεταξύ 5 και 11% του ΑΕΠ. Και μάλιστα το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά λόγω των δημογραφικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική ευθύνη, χρειαζόμαστε αξιόπιστους δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι και να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται και να ενισχυθούν μάλιστα για να ολοκληρωθεί επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των οικονομικών, των δημοσιονομικών μάλλον δαπανών πρέπει επίση να είναι εξασφαλισμένη και αυτή όμως θα αλλάξει λόγω των δημογραφικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν δείκτη που θα επιτρέπει την αξιολόγηση σε ποιο βαθμό οι εθνικοί προϋπολογισμοί επηρεάζουν τις μελλοντικές γενιές. Και τέλος, Η δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία πρέπει να βελτιωθεί. Οι εθνικές βουλές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαλέγονται καλύτερα ε, στη βάση συστάσεων αναχώρα. Οι οποίες συστάσεις αναχώρα θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές αυτή τη στιγμή τις υιοθετούν επισήμως οι κυβερνήσεις. Και αναμένω τις συνεργασίες μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Μου φαίνεται ότι δεν είναι εδώ κανείς από την Ενωτική Αριστερά, ούτε και από τους Πράσινους, ούτε και από την ομάδα EFDD. Τώρα η ομάδα ENF. Εσείς, κυρία μου, για το λογαριασμό του EFDD, όχι. Καλά, εσείς τότε για το, την Ευρώπη των Εθνών. Ο κύριος Άνεμανς. Ευχαριστώ. Θα κοιτάξω εννοείται πολύ προσεκτικά όταν θα έχουμε το τελικό κείμενο. Συνήθως όλες αυτές ε, οι εκθέσεις αποτελούν μέρος ενός συνόλου που έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και πρέπει να κοιτάμε και πάρα έξω έτσι ώστε να εμπνεόμαστε για το τι πρέπει να κάνουμε με ελεύθερη αγορά, τι έφερε το Μάστριχτ, να κάνουμε αξιολόγηση, να δούμε τι πρέπει να στηρίξουμε και τι δεν πήγε καλά. Ποιες είναι οι επιπτώσεις επίσης του ενιαίου νομίσματος που μερικές φορές ήταν καταστροφικές για την οικονομική ανάπτυξη και δεν πρέπει να τα παρατείνουμε αυτά είναι θέμα ταυτότητας, ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης που έχουν επιπτώσεις και στον οικονομικό τομέα, στην οικονομική δύναμη της Ευρώπης. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα άλλο μοντέλο και να μην συνεχίζουμε την πολιτική μας όπως μέχρι τώρα. Έχουμε παγιδευτεί. Το σύστημα αυτό όσο δεν το αναφερούμε και δεν το αλλάζουμε θα παραμένουμε παγιδευμένοι σε αυτό. Αυτά που παρουσιάζει ο κύριος Χόμαρ μπορεί να μην το συνειδητοποιεί, αλλά ουσιαστικά παραμένει στο ίδιο σύστημα. Προτείνει κάποια μικρή ανάπτυξη με τα μέτρα αυτά, αλλά πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές αν θέλουμε όντω να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό που είπε για τα πόδια στο φούρνο και το κεφάλι ε, στο ψυγείο έχει δίκιο. Δεν είναι ο μέσος όρος που πρέπει να μας καθοδηγεί πάντα. Πρέπει να είμαστε επικριτικοί όπως είμαστε και εμείς απέναντι στην έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. ΆΗ. η Υπερβάνος Μπερές έχει ζητήσει το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και μετά και ο κύριος Ροζάτη. Είναι πρώτος μήπω ο κύριος Ροζέτη. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Εισάγει μια νέα έννοια, αυτή του ψυγείου και του φούρνου που λέγαμε. για να εξηγήσει πως έχουμε μια πόλωση στα οικονομικά ζητήματα. Τα διδάγματα αυτά όμως δεν τα χρησιμοποιεί ο ίδιος ε, στα συμπεράσματά του, γιατί μας λέει ότι υπήρξαν κίνητρα στήριξη δημοσιονομική, αλλά όσον αφορά τις αλλαγές δεν έχουν γίνει αρκετές. Όμως ένα από τα πράγματα τα οποία ακριβώ χαρακτηρίζουν την πολιτική συζήτηση σήμερα είναι η κόποση που διαπιστώνουμε σε μερικές χώρες μέλη. Δεν είναι τόσο ότι υπήρξαν ε, πολλά οικονομικά κίνητρα, γιατί τότε δεν θα χρειαζόμασταν το σχέδιο Juncker, αλλά είναι η πρακτική των διαρθρωτικών αλλαγών, έτσι όπως την αντιληφθήκαμε στην πρώτη γενιά, που ήταν προσανατολισμένη στη μείωση του κόστους και άρα ανταγωνιστικότητα στο κόστος. Εγώ προτείνω να βγούμε από αυτή την πόλωση, ψυγείο και φούρνος, για να συνοδεύσουμε διορθωτικές αλλαγές νέας γενιάς. Να γίνει συζήτηση για κίνητρα προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, ζώνη ευρώ ιδιαίτερα. Ο κύριος Ροζάτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Χόκμαρ για την τόσο καλή του έκθεση συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις του και τις συστάσεις του. Έχω την άποψη ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δαπανών καλύτερο και φυσικά να λάβουμε υπόψη μας τις επενδύσεις, κυρίως τις υποδομές. Και αυτό πρέπει να αναφέρεται στην αρχή του καταλόγου για τις δαπάνες μας. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε εξαιρέσει, κάθε φορά που δημιουργούμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες κατηγορίες δαπανών που να ξεπερνούν το όριο, τότε η κατηγορία αυτή βγαίνει από τις τακτικές δαπάνες. Βάζουμε όλα τα υπόλοιπα στις τακτικές ε, δαπάνες, ξέροντας ότι οι έκτακτες μπορούν πάντα να είναι εκτός ορίου. Δεν είναι καλή προσέγγιση αυτή. Δεύτερον, για τα δημοσιονομικά κίνητρα. Ο κύριος Χόκμαρ λέει ότι υπάρχουν πολλά τέτοια στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι έχει στο μυαλό του τα επίπεδα ε, χρέους. Όντως υπήρξαν δημοσιονομικές ε, δαπάνες, οι οποίες όμως δεν πήγαιναν εκεί που θα έπρεπε να πάνε. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Άλλε χώρε έχουν δημοσιονομικά περιθώρια και μπορούν να δαπανίσουν παραπάνω. Αλλά η αύξηση των δημοσιονομικών ε, δαπανών και η ενίσχυση της οικονομίας τους είναι δικό τους θέμα. Δεν είμαστε εμείς που πρέπει να τους πούμε στη Γερμανία, στις κάτω χώρες Δεν υπάρχει μέσο για να πείσουμε τις χώρες αυτές να δαπανίσουν περισσότερο. Αν επιθυμούν να δαπανίσουν περισσότερα θα το κάνουν. Αν δεν θέλουν όμως δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε. Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες που είναι υπερχρεωμένες και δεν έχουν τέτοιο δημοσιονομικό περιθώριο. Οπότε σε τι βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές ε, τις χώρες από τις συνολικές δαπάνες στην Ευρωζώνη, όσο δεν διαθέτουμε τα πολιτικά εργαλεία, τα οποία με κάποιο τρόπο θα βάλουν σε μη δημοσιονομική πολιτική όλη την δημοσιονομική κυριαρχία των χωρών μελών, δεν μπορούμε να ελπίσουμε τίποτα άλλο. Επίσης, για αυτά που είπε ο κύριος Λούκατς πριν, συμφωνώ για αυτά που είπε για την ανταγωνιστικότητα και για τις αιτίε έλλειψης επενδύσεων στην Ευρώπη. Το πρόβλημά μου όμως είναι η αξιολόγησή του όσον αφορά το ρόλο που έχει παίξει το ευρώ και αυτό το λέω και για τον άλλο συνάδελφο που αναφέρθηκε στην Ευρωζώνη. Αν ο κύριο Λούκατ πιστεύει ότι οι χώρε αυτέ με δικό του νόμισμα, με υποτίμησή του, θα είχαν μπορέσει να διορθώσουν την κατάσταση, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια αυτή. Όταν υποτιμά το νόμισμά σου, δεν γίνεσαι πιο ανταγωνιστικό και γίνεσαι πιο φτηνό. Δεν γίνεσαι πιο καινοτόμο, πιο παραγωγικό, πιο φθηνό γίνεσαι μόνο. Μακροπρόθεσμα αυτό δεν είναι λύση. Σαν να κουφίζει βραχυπρόθεσμα, αλλά τίποτα άλλο μετά. Ευχαριστούμε. Φίλιπ Λάμπερς τώρα. Θέλω να αντιδράσω σε αυτά που μόλι τώρα είπε ο κύριο Ρωσάτη. συμφωνώ με το τελευταίο που είπε. Δεν είναι επειδή γίνεσαι πιο φθηνό που γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός. Σωστό, γιατί η πραγματική ανταγωνιστικότητα προέρχεται από την διάθεση αγαθών και προϊόντων που προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Αυτή είναι η πραγματική ανταγωνιστικότητα, η σκληρή ανταγωνιστικότητα. Αλλιώς ε, είναι αυτινός τρόπος και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω και το ξαναλέω και μου αρέσει αυτό που είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να μην βασιστεί ε, στο χαμηλό κόστος. Δεν είμαστε μια ήπειρος χαμηλού κόστους, αντίθετα στο ψηλό κόστος. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα με τα οποία θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στις χώρες που από μόνες τους δεν μπορούν να έχουν επενδύσεις. Υπάρχει ένα έμεσο μέσο. Αν δείτε το six packs και τη διαδικασία μακροοικονομικών ισορροπιών, εκεί έχουμε έναν έμεσο τρόπο προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στις χώρες να επενδύσουν. Όταν έχετε υπερβολικό πλεόνεσμα και τότε επιμέναμε να συμπεριληφθεί αυτό στην νομοθεσία και η Κομισιόν κάνει σαν να μην υπάρχει αυτό. Πάντως όταν υπάρχουν τέτοια μαζικά πλεονάσματα αυτά τι σημαίνουν. ότι μια χώρα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αλλά μπορούμε να το δούμε κι αλλιώς, σαν ένα δείγμα έλλειψης κατανάλωσης, υποκατανάλωσης. Όταν τα βάζουμε με τη Γερμανία, επειδή έχει τόσο μεγάλα πλονάσματα, δεν είναι επειδή μπορεί και τα εξάγει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τέχνητα περιορίζει την εσωτερική ζήτηση η Γερμανία. Θα προτιμούσαμε λοιπόν επενδύσεις από την ε, κατανάλωση, εννοείται ότι χρειάζεται και η κατανάλωση, αλλά την οικονομία σας μην την κινείτε και πάλι βάση της κατανάλωσης μόνο. Χρειάζονται και επενδύσεις. Μου φαίνεται ανόητο το σχέδιο Juncker να χρηματοδοτεί επενδύσεις στη Γερμανία όταν η Γερμανία έχει τεράστιες δυνατότητες επενδυτικές. Αυτό είναι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα έμεσο εργαλείο, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι καλό και καταγγέλλω το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το χρησιμοποιεί. Ο κύριο Λούκα μου είπε ότι ένα λεπτό μόνο θα αντιδράσει. Παρακαλώ. Ο κύριο Λούκα, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφους μου, η FDD και αριστερά που επιτρέπουν να γίνει και κάποια συζήτηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Λάμπερτ, ο οποίο αμφισβητεί τον ισχυρισμό μου, αλλά στην ουσία τον επιβεβαιώνει, λέγοντα ότι ε, ο ανταγωνισμός γίνεται σε δύο επίπεδα. Μπορεί δηλαδή και στην αξία, στο επίπεδο της αξίας και στο επίπεδο του κόστους. Βεβαίως, ο ανταγωνισμός ενισχύεται και όταν μειώνεις τις τιμές. Αν είσαι χαμηλότερες τιμές, είσαι πιο ανταγωνιστικός. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο σκέλη. Αν όμως η διαφορά των τιμών είναι τόσο τεράστια, όπως συμβαίνει τώρα στην Ευρωζώνη, όπου οι υποτιμήσεις είναι σημαντικές και φτάνουν στο 30-40% για ορισμένε χώρε τη Ευρωζώνη. Είναι απολύτω μη ρεαλιστικό να αναμένει κανεί ότι οι επιχειρήσει σε αυτέ τι χώρε τη κρίσεω θα μπορέσουν να επιτύχουν κέρδη σε ό,τι αφορά την ποιότητα του προϊόντο που να καλύψουν το 40% διαφορά των τιμών του. Αυτό που χρειάζονται λοιπόν αυτέ οι επιχειρήσει είναι πρώτον υποτίμηση, χαμηλότερε δηλαδή τιμέ, έτσι ώστε να αρχίσει να αποδίδει η επένδυση σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα, είναι σαφές, λοιπόν το, το νόημά σας, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ που μου δώσατε χρόνο. Πρέπει να υπάρχει και κάποια ευκαμψία και στην ε, χορήγηση χρόνου ε, στο κάτσε Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δεν θα επανέλθω σε όλα. Πρώτα, ωστόσο, νομίζω ότι σωστό είναι να γινόμαστε ανταγωνιστές με υψηλές αμοιβέ. Βεβαίω πάντα μπορεί να χαμηλώσει κανεί τι τιμέ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλύτερε δουλειέ. Αυτό που προκύπτει από τη συζήτηση πάντω νομίζω ότι είναι. Είναι ότι δεν αμφισβητείται τουλάχιστον τι μεγάλε πολιτικέ ομάδε το σύμφωνο σταθερότητο. μάλιστα το ερμηνεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο ότι η συζήτηση για την θετική δημοσιονομική στάση δεν υπονομεύει τη σταθερότητα του, το μάλλον την αξία του θεσμού Σταθερότητα και την αξιοπιστία του. Θα επανέλθω τώρα στο μαγειρίο μου για να σας ε, ξαναμιλήσω για ε, ψυγεία και φούρνους, γιατί είναι σημαντικό για μας να αντιληφθούμε ότι οι διαφορετικές χώρες μέλη εξελίσσονται διαφορετικά. Είπαν ότι έχουμε έλλειψη ανάπτυξης. Σωστό. Συνολικά. Γιατί υπάρχει και σε ορισμένε άλλε χώρε μέλη ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και υψηλό επίπεδο επενδύσεων. Και αυτό συχνά συνδέεται και με τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Έχουμε μια εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και καμιά φορά εκεί αυτό έρχεται σε αντίθεση, σε αντίφαση μάλλον. γιατί σε ορισμένες χώρες έχουμε εκεί μάλλον και το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτές τις αποστάσεις, τις αποκλήσεις. Ίσως η λύση να μην είναι πάντοτε η αύξηση του χρέους. Ίσως για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα να είναι το πιο σημαντικό οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις. Χωρίς να έρχομαι σε αντίφαση με αυτό που είπατε εσείς, Περβάμος, ότι χρειάζονται και δημόσιες επενδύσεις για να ενισχυθούν οι οικονομικοί δείκτες. Τα και άλλα, και άλλα αυτά. Θα τα περιλάβω αυτά. Άλλωστε αντιλήφθην και μια προθυμία για να καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, προτάσεις. Θα συζητήσω και περαιτέρω βεβαίω με τους ηγητέ και με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη θετική σας στάση απέναντι στους ε, συμβιβασμούς. Αναμένουμε την εργασία σας. Βεβαίως το σύμφωνο σταθερότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρως και με την ευελιξία που ε, περιλαμβάνεται άλλωστε μέσα στο ίδιο σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα εξευρεθούν λογικές συμβαστικές ε, λύσεις στις ε, διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει. 6 Φεβρουαρίου και ελπίζω στην Ολομέλεια 13 Φεβρουαρίου. Το επόμενο τώρα της ημερησίας διατάξεως του κυρίου Λάμπερτς η έκθεση για την καθίδρυση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την στήριξη της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών ε, υπηρεσιών για την ε, συμμετοχή τους λοιπόν στην περίοδο 2017 έως 20. Παραδίδω και τα ενία της ε, συζητήσεως στον κύριο Φέρμπερ. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως θα έχετε διαβάσει από τις συμβαστικές τροπολογίες, προσπαθήσαμε να περιλάβουμε όλε τι απόψει, όλων όσοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Ορισμένοι εξημών δεν το ε, υποστηρίζετε, αλλά οι περισσότεροι το υποστηρίζετε. Και μάλιστα προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και τα όσα μα ήλθαν εκ τη ΙΜΚΟ, ιδίω για την 6 και 7 εκεί η, η Επιτροπή αυτή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και αλλού έχουμε κοινή αρμοδιότητα. Με λίγα λόγια, δεν απέχει πολύ η πρότασή μου από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Θα περάσω λοιπόν τα διάφορα άρθρα ε, σχετικά γρήγορα. Άρθρο πρώτο, δραστηριότητες, εκεί περιλαμβάνουμε, οι οποίες χρηματοδοτούνται δηλαδή, και ε, με του ε, δημοσίου συμφέροντος. Και για την εμπλοκή δικτύων καταναλωτών. Στο δεύτερο αυτό τώρα στον χώρο των δημοσιονομικών κανονισμών το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει και τους τελικούς χρήστες όχι μόνο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα όπως για παράδειγμα το πολυμερές. Έχουμε και την τροπολογία της ΙΜΚΟ 25 για τις νομισματικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους δικαιούχους του προγράμματος. Άρθρο 3 για τους δικαιούχους Εκεί έχει προταθεί από πολλούς και από την ΙΜΚΟ οι δικαιώχοι του προγράμματος να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους μέσα στις ίδιες τις χώρες μέλη ώστε να μην παραμείνει μέσα στο κέλυφος, το κλειστό κέλυφος των Βρυξελών, αλλά να μπορέσει να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες μέλη. Δεν έχουμε σημαντικές τροπολογίες για το 7, εφαρμογή του προγράμματος. Αποφασίσαμε λοιπόν να δεχθούμε το κείμενο της ΙΜΚΟ. 9. Αξιολόγηση. Σύρπα και Ενρίκη έχουν κάνει προτάσει εκεί. για να ανατεθεί και σε άλλε οργανώσει εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα και σε νέα περίοδο. Η αξιολόγηση της Κομισιόν θα εξετάζει και το ενδεχόμενο να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος. Με άλλα λόγια, κοιτάμε την επόμενη περίοδο με ανοιχτό πνεύμα και σε ό,τι αφορά τους ενδεχόμενου δικαιούχου αλλά και σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά ποσά. Μετά δε, από συζήτηση και με τις υπηρεσίε κομισιών αλλά και με τους μελλοντικούς δικαιούχους, απολογία για το άρθρο 10 που λέει ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαΐου 2017 και θα πάει μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου 2020 για να ε, χρηματοδοτηθούν οι δικαιούχοι και έχοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις αρχίζουν από τις 30 Απριλίου. Δεν θέλουμε δε να υπάρχει οικονομικό κενό ανάμεσα στο τέλος του ενός προγράμματος και στην αρχή του επομένου. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, μια στιγμή να βρω τις ε, σημειώσεις μου, ο σχεδιασμός μας είναι γραπτή διαδικασία, θα σας στείλουμε δεύτερο σετ, δεύτερο σύνολο ε, συμβαστικών τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 25 πρώτου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αμφιγνωμία μεταξύ μόνο και του Συμβουλίου, άρα θα μπορέσουμε έγκαιρα να το εγκρίνουμε στην Ολομέλεια, ώστε να μην υπάρξει αυτό το χρηματοδοτικό κενό. Ευχαριστώ, λέω ο Προεδρεύων Φέρβερ. Παρακαλώ, οι ο δε κύριος Στόλογιαν εκπροσωπεί την κυρία Πιετικάινεν για λογαριασμό του Λαϊκού κόμματο όλα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Πιετικάινεν υπέβαλε έναν σχετικό αριθμό τροπολογιών στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να αναφερθούν οι δύο δικαιούχοι του προγράμματος ε, στον κανονισμό ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία των δύο αυτών οργανισμών προ όφελο όλων. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται καθυστερημένα ε, με την ανάγκη χρηματοδότηση να αρχίσει ήδη από την αρχή τη χρονιά και δυσκολεύει και τους ετούντες και τη λειτουργία των δύο οργανισμών ε, για το 2017, βάζοντα σε κίνδυνο την ε, εύρυθμη λειτουργία τους. Δεν υπάρχει άλλος οργανισμός που θα μπορούσε να καλύψει τις ίδιες ε, αρμοδιότητες και ανάγκες. Και αυτό το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Πιτικάιναν λοιπόν θα ήθελε να ότι το πιλωτικό πρόγραμμα και η σχετική χρηματοδότηση που είχε προβλεφθεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην διακομματική ε, έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίση, ζητά η χρηματοδότηση να ξεπεράσει το προβλεπόμενο τώρα διάστημα 2017-2020 και στο μέλλον η προκήρυξη να είναι ανοιχτή σε όλους τους ε, δεχόμενους ε, δικαιούχους εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Θα ήθελε η λειτουργία των δύο οργανισμών αυτό το διάστημα να ε, καλύψει γεωγραφικά περισσότερα κάτι μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλε Λούντβιξον, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Η ερώτηση είναι εάν μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χρειαζόμαστε στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδότηση και πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει η τεχνικότερη νομοθεσία να γίνει κατανοητή για τους καταναλωτές. Επίσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η λειτουργία των οργανισμών αυτών είναι εξαρτητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαρτάται η εμπιστοσύνη του κοινού από αυτό το στοιχείο. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη στη λειτουργία του από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα. Μακροπρόθεσμα είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ε, οικονομική τους ανεξαρτησία επίσης. Και οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν θα είναι απλός ο δρόμος. Οι οργανισμοί αυτοί θέλουν να είναι ανεξάρτητοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλά δικαιώματα παρακολούθησης και επίβλεψης των δύο φορέων. Ενδεχομένως να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων ως προς την ανεξαρτησία των δύο θεσμικών αυτών οργάνων. Και οι χρηματοοικονομικοί τους πόροι είναι περιορισμένοι. Δεν μπορούν να κάνουν και τα πάντα σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα δίκτυα και οι ενεργοί φορεί στα διαφορετικά τη κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, και αυτό το ρόλο του που θα είναι σημαντικό στο μέλλον. Είμαι βέβαιο ότι σε συνεργασία με τον εισηγητή και του υπολείπου σκιώδη θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλοι. Και τώρα για τους φιλελεύθερους ο κύριος Ντεσάμπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύντομα, λοιπόν. Η ομάδα μου θα τοποθετηθεί υπέρ του κειμένου της Επιτροπής και των τροπολογιών που με ξέρετο τρόπο συνέλεξε ο συνάδελφος Λάμπερτ. Διαβάσαμε τις συμβαστικές προτάσεις, πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, οπότε θα τα καταφέρουμε. Το πρόβλημα που μπορεί να τεθεί είναι πολιτικής φύσης. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κάποιο τρόπο καταπίνει την επιτυχία της πρότασής μας. Οι ομάδες μελέτης δεν πρέπει να θεωρούν ότι εκείνες εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Εμείς εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ δεν ξεχνώ ποτέ τις υποχρεώσεις μου και δεν θα ήθελα ούτε και οι συνάδελφοι να τις ξεχνάνε. Οι ομάδες αυτές υπάρχουν για να βοηθούν τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου η εκτελεστική εξουσία να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Στη γραμμή όμως που λέει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όχι να προσπαθούν να πάνε κατά των όσων λένε οι άλλοι, αντίθετα να ενισχύουν αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, συμφωνώ και πιστεύω ότι με το κύρος του συγκητή και του κοινοβουλίου μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Κανένας βέβαια δεν πρέπει να είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Όπως λέει και ο κύριος Λάμπερ, πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όχι μόνο τους καταναλωτές, τους τελικούς επενδυτές, όσους παίρνουν αποφάσεις, όχι μόνο στις Βρυξέλλες και αλλού. Πρέπει να αποτελεί μια δημόσια υπηρεσία, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάνε πολλές τροπολογίες. Τέλος, για να μην υπάρχουν υπόνοιες, οι δύο οργανώσεις Better Finance και Finance Watch έχουν το πλεονέκτημα ότι τις έχουμε υποδεχτεί ιδιαίτερα θετικά. Όμως πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε στο μέλλον εξακολουθούν να είναι οι κατάλληλες και να μην υπάρχει υπόνοια ότι το Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή χρηματοδοτούν. Με την τροπολογία πάντως επίσης του κύριου Λαμπέρτ νομίζω ότι το πετυχαίνουμε αυτό γιατί λέω ότι θα είναι ανοιχτέ και καλύτερα χρηματοδοτούμενε. Λοιπόν, το πολιτικό ζήτημα μένει γιατί τα τεχνικά ζητήματα έχουν λυθεί πλήρως από το κείμενο της Κομισιόν και της τροπολογίας της ΣΥΜΚΟ και του κύριου Λάμπερτς. Συνεπώς πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την κοινωνία των πολιτών που εμείς εδώ εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Με κάθε τώρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή, το σχέδιο έκθεσης και τις συμβαστικές τροπολογίες που πήραμε οι σκιώδες στις αρχές της εβδομάδας. Αν εγκριθούν οι συμβαστικέ τροπολογίε από το Κοινοβούλιο, βελτιώνεται σημαντικά η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί θέλουμε να αναγνωρίζετε ότι το έργο τη Finance Watch και τη ε, Better Finance είναι σε πλαίσια συμβουλών για καλύτερη πολιτική από πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Είναι πολύτιμε συμβουλέ. Οι οργανώσει αυτέ έχουν ένα ρόλο να παίξουν όχι μόνο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και γενικότερα σε κάθε περίπτωση λήψης πολιτικών αποφάσεων από άλλα φόρα. Πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τον ρόλο των οργανώσεων αυτών για να ακολουθούμε θεμητές οικονομικές πρακτικές. Όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα, θέλουμε οργανώσεις αυτές να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό ζητούμε οι ομάδες που ασχολούμαστε με τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ε, στηρίζουμε και την πρόταση που λέει ότι οι οργανώσεις αυτές πρέπει να περιγράφουν το σχέδιο δραστηριοτήτων τους και την πρόταση του συγητή και του MCO που λένε ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για, την καλύτερη, για τα καλύτερα οικονομικά χρηματοδότηση κτλ. Στις συμβαστικέ προτάσεις αναφέρεται και η έμεση χρηματοδότηση. Λοιπόν, συμφωνούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρόεδρε, εγώ ευχαριστούμε πολύ. Έξω από το EFTD. Ευχαριστώ. Όπως είδατε, αλλά και ε, όπως θα αντιληφθείτε, δεν μπορώ να στηρίξω την πρόταση αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πρόκειται για χρηματοδότηση από ε, χρήμα των φορολογουμένων και μάλιστα σε ύψη πολλών εκατομμυρίων. Και στην ουσία πρόκειται για λόμπι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Και υπάρχει ένα παράδοξο, αν το καλοσκεφτούμε. Πάμε να στηρίξουμε μια, ένα λόμπι με χρηματοδότηση πολλών εκατομμυρίων. Γιατί να μην χρηματοδοτήσουμε τους καταναλωτές χωρίς το λόμπι αυτό. Για δέστε και ποια είναι τα μέλη της Finance Watch. Είναι η Attack France, το Ίδρυμα Heinrich Böll των Πράσινων, ή το Ίδρυμα Ρώσα Λούξεμπουργκ των Αριστερών. Ρωτώ λοιπόν τους συντηρητικούς συναδέλφους μου, σας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Πάτε να διαθέσετε χρήμα των φορολογουμένων σας σε αυτά τα κανάλια. Εγώ δεν συμφωνώ. Έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Μακάρι να το κάνετε. Εγώ θα το κάνω και θα απορρίψω την πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Φέρμπερ. Από το ΙΝΕΦ. όχι. Δεν έχουμε κάτι the για την ώρα τουλάχιστον. Ο εισηγητή λοιπόν. Ε, νομίζω ότι όντω διαμορφώνεται μια ευρεία συνένεση ανάμεσα σε αρκετά κόμματα για να περάσει η πρόταση. Αναμένω τα σχόλιά σα για το πρώτο σύνολο συμβαστικών τροπολογιών το συντομότερο δυνατό ώστε να μπορέσω να τα περιλάβω και να συνεχίσω για την κυρία Φων Στόρκ σας έχω απαντήσει και άλλες φορές. Ίσως αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται για κερδοσκοπικές οργανώσεις. Όταν μιλείτε για λόμπι, τα λόμπι στηρίζουν κερδοσκοπικές οργανώσεις. Κανείς δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά εδώ. Το μόνο κέρδος που θα αποκομίσουν είναι οι καταναλωτές. Ναι, λέτε ότι στηρίζουμε τους καταναλωτές με, με... με χρήματα φορολογουμένων. Εν μέρει ναι. Όμως όπως γνωρίζετε κάθε καλή δημοσιονομική ρύθμιση αποδίδει υπέρ των καταναλωτών. Διότι αν δεν τα κάνουμε αυτά, ποιοι τα πληρώνουν τελικά, οι φορολογούμενοι. Και δεν πάμε πλέον να μιλήσουμε για ορισμένα εκατομμύρια, μιλούμε για δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν οι φορολογούμενοι επειδή οι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν εποπτεύονταν ορθά. Το να ξοδέψουμε λίγα λοιπόν εκατομμύρια για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από αυτούς που δεν κάνουν στα τα πράγματα, ε, είναι λοιπόν σωστά δαπανημένα. Γνωρίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει να υποστηρίζετε τους καταναλωτές, σας ενδιαφέρει περισσότερο να ενισχύετε τον ιδιωτικό κλάδο, τη ιδιωτική βιομηχανία και όσους απολαμβάνουν από αυτήν. Αυτές είναι οι διαφορές μας. κανείς δεν εκπροσωπεί καλύτερα, επιτρέψτε μου την προσωπική αυτή παρατήρηση, του τους Ευρωπαίους από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσωπική παρατήρηση αυτή, όχι ω Πρόεδρο. Θα ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου και τον Μάρτιο πλέον στην Ολομέλεια. Έχω τώρα τα υπαριθμών 6, 7 και 8. Πρόκειται για την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών. Σάντερ Λούνς. Σάντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το δώρο μου για την καινούργια χρονιά είναι αυτή η απαλλαγή, η τριπλή απαλλαγή και οι σχετικές νομοδοτήσεις. Όπως ξέρετε είχαμε πολύ μεγάλη χρονική πίεση και, ε, και περιορισμό στην έκταση των νομοδοτήσεων Υπήρξαν και αρκετέ τροπολογίε. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Θα επικεντρωθώ σε τρει βασικέ παρατηρήσει. Πρώτον, κατά την άποψή μου, και αυτό αναφέρεται και στι νομοδοτήσει, δεν θα πρέπει το πεδίο νομοδοτήτων των ε, αρχών αυτών να διευρυνθεί. Θα πρέπει να παραμείνει και επιχειριστή στην αρχή και να δώσουμε και προσοχή στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην περίπτωσή τους. Πιστεύω ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος. Θα ήθελα όμως και τη γνώμη των σκοτών ψηφιτών. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει αυτές οι αρχές να χρησιμοποιούν τον προπολογισμό τους με τρόπο χρηστό, δηλαδή οποιασδήποτε επιπλέον επίσης για πόρους θα πρέπει να δικαιολογούνται και να συνοδεύονται από μέτρα εξωτερικισμού. Λόγου χάρη αλλάζει αρκετά η δουλειά των αρχών αυτών από την ομοθετική δουλειά προς την ε, ε, παρακολούθηση της σύγκλησης και την υλοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσαρμοστεί και ο προπλογισμός τους και η επάντρωσή τους. Και τέλος αναφέρουμε και την επερχόμενη αναθεώρηση των οικονομικών διευθετήσεων ε, για τις αρχές αυτές. Θα δείτε και το σχετικό οικονομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πότε θα προκύψει η Λευκή Βίβλος της ευρωπαϊκή επιτροπή για τις ε, Ευρωπαϊκές Αρχές και την ε, οικονομική του διακυβέρνηση, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι το κείμενο αυτό θα προκαλέσει σωρία συζητήσεων όχι μόνο στον χώρο των οικονομολόγων και των χρηματοπιστωτικών ειδημόνων αλλά και στο επίπεδο των πολιτικών εθνόντων. Περιμένω λοιπόν με τα χαρά στα σχόλια και τις τροπολογίες σας. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε ευρεία πλειοψηφία και στις τρεις περιπτώσεις. Σε ευχαριστούμε, Ζάντερ. Δεν έχει φτάσει ο συγκεκριτή μα από το ΕΛΚ, είναι στη διάσκεψη των Πρόεδρων, οπότε θα αλλάξω τη σειρά των ομιλητών και πρώτοι θα πάρουν το λόγο σοσιαλιστέ. Ο Σόρου Φρουντζουλίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τη γνωμότησή του για τις απαλλαγές του 2015 για τις τρεις ευρωπαϊκές αρχές. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντική η ετήσια απαλλαγή ως μέτρο να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα και να επιφέρουμε διορθώσεις. Και η ΕΟΠΑ και η ΕΠΑ και η ΑΤ και η ΕΣΜΑ έχουν στόχο να προσφέρουν συστημική σταθερότητα και προστασία των ε, πολιτών και επειδή ε, πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμό στον προπολογισμό τους ε, και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πληρώνουν το λογαριασμό οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Ε, θα πρέπει οι συγκεκριμένες αρχέ να ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους και την δράση τους. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στη δουλειά τους προκειμένου οι, οι μέρημνες και δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να την χάνουν σωστή μεταχείριση. Και η οικονομική σταθερότητα θα πρέπει να παραμείνει ο βασικό στόχο λειτουργία αυτών των αρχών. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι η ΙΟΠΑ θα πρέπει να παρακολουθείτε σωστά ε, και να παρακολουθεί τι συμβαίνει όταν οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν λειτουργούν αρκετά ε, σωστά. Ε, για να βεβαιώνει τη σωστή λειτουργία των ε, αγορών, όπως συνέβη με τη Ρουμανική Αρχή για την αγορά της Ρουμανίας το 2015. Ίσως ξέρετε ότι το Ρουμανικό Κοινοβούλιο ε, εκείνησε διαδικασία για να απολυθεί ο πρόεδρος της Ρουμανικής Εθνικής Εποπτικής Αρχής λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί. Σε ό,τι αφορά την ΕΜΠΑ, την Αρχή των Τραπεζών. θα πρέπει να αναθεωρηθεί η λειτουργία της στο πλαίσιο και της Τραπεζικής Ένωσης. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή, η κάθε Ευρωπαϊκή Αρχή, να, ενημερώ, να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί τις πληροφορίε σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων τη και τη δράση της και να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας για την δουλειά και την πρόοδο που ε, επιτελείται θέλουμε να φτάσουμε ε, στο ευρύτερο κοινό, ενδεχομένως και μέσω web streaming. Είμαι πρόθυμος να ε, συνεργαστώ με τους υπόλοιπους συναδέλφους για να βρούμε τις σωστές τροπολογίες, βεβαίως με τον ίδιο τον εισηγητή, και να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Πάλι δεν έχει φτάσει ο εισηγητής ε, του ΕΛΚ. Από τους φιλελευθέρους δεν βλέπω κανέναν. Από τους πρασίνους. Φίλιπ. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο. Μέρος της εκτίμησής του το συμμεριζόμαστε. ιδίω την ανάγκη να αναθεωρηθούν κάποιες οικονομικές διευθυντήσεις με την εισαγωγή αναλόγων τελών, κατάλληλων τελών για τους συμμετέχοντες στην αγορά και με τη συμβολή των εθνικών εποπτικών αρχών και τη βελτίωση της ποιότητας και της ε, συνολικής κάλυψης με την παραγωγή των πρακτικών λειτουργίας των αρχών. Βέβαια είναι κάπως περιοριστική η προσέγγιση των τριών γνωμοδοτήσεων ως προς τον προβλαγισμό που θα προβλεφθεί για τις αρχές αυτές. Ξέρετε ότι από τη στιγμή που ιδρύθηκαν αυτές οι αρχές, στον αντίκτυπο της κρίσης, διαρκώς συνηγορούσαμε υπέρ της αύξησης των, αρχών, των πόρων που θα τους ε, δίδονται. Και στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι θα κάνουμε ως προς την διάθεση πόρων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει διαφάνεια και ανεξαρτησία, αλλά θέλουμε και οι ευρωπαϊκέ αρχέ να προβλέψουν ένα ασφαλή διάβλο για να προστατεύονται και οι πληροφοριοδότε, οι whistleblowers. Και θα πρέπει τα διάφορα έγγραφα που ε, σχετίζονται με τι διάφορε υποθέσει που εξετάζουν οι αρχέ να δίδονται και στου ενδιαφερόμενου όπω το Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότεροι πόροι για την σωστή υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου και την προστασία των καταναλωτών. Οι αρχέ δεν έχουν ακόμα εξασκήσει όλε τι αρμοδιότητε που του έχουν ε, αποδοθεί, όπω την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, την προστασία των καταναλωτών, τι ε, εκθέσει ε, ομοτήμων και ούτω Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούν όλε τι δυνατότητε που του δίνει η νομοθεσία και γι' αυτό έχουμε υποβάλει τροπολογίε για να απηχηθεί και αυτή η άποψη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λάγκεν βλέπω ότι φτάνει ε, ο Μάρκο Βάλλη. Η ευθυντή και άλλη Α, κύριε Άνεμαντς. Ναι, η κυρία Κάπελ δεν ε, μπορεί να είναι εδώ. Εγώ δεν θέλω να αναιρέσω το έργο του κύριου Λόνης καθ' άλλο, αλλά Πέρυσι, το 2015, ο κύριος Μάρκους Φέμπερ είχε τις ε, εκθέσεις και χαιρετίζω για την ΕΣΜΑ, για ότι τα αποτελέσματα θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται, να προβληθεί αυτό. Για τα άλλα δύο, είπαμε και πέρυσι ότι οι φιλοδοξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν πολύ νόημα. Μιλούσαμε για έναν ευρύτερο ρόλο ήδη από πέρυσι. Market Participants για την ΙΟΠΑ, ε, την ε, Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών ότι πρέπει να υπάρχει μια στάθμιση για να μην είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Ελπίζω, θα εισηγήσουμε τέλο πάντων εμείς τα πράγματα για να δούμε ανάλογα με τις τροπολογίες αν μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά που δεν βρίσκουμε καλά. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα που να εκπλήσει. Ευχαριστούμε. Τώρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν ήμουν στην ώρα μου σήμερα. Θα έπρεπε να είχα οργανωθεί καλύτερα. Τέλος πάντων. Ομολογώ ότι κάπω απογοητεύτηκα, ομολογώ, από την οξύτητα των ε, όσων έγραψε το λεκτικό συνέδριο. Δεν βλέπω τίποτα ενδιαφέρον. Φυσικά αναφέρονται τα καθήκοντα, αλλά τελικά δεν μαθαίνουμε και πολλά από τις εκθέσεις αυτές. Απογοητεύτηκα λοιπόν και αναρωτιέμαι, μήπω στο μέλλον θα έπρεπε να ζητάμε από, την εκθε... από το ελεκτικό συνέδριο να μα παρουσιάζει πιο λεπτομερεί εκθέσει. Δεύτερον, όντω το 2011 ήμουνα εγώ για δύο από αυτές τις τρεις απαλλαγέ εισηγητή. Τότε η κατάσταση ήταν βέβαια πολύ διαφορετική σε σχέση με σήμερα. Ε, πάλι δεν είχαν λειτουργήσει όλα καλά, τα είχε εντοπίσει το ελεκτικό συνέδριο και τα τελευταία χρόνια Ρόλος μας ήταν η βελτίωση αυτών των σημείων, να διορθωθούν κάποια πράγματα. Υπήρξαν εκθέσεις από το Ελληνικό Συνέδριο που έλεγαν ότι σιγά σιγά προχωράμε, σιγά σιγά, βήμα βήμα. Αξιολογούμε λοιπόν το έργο και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί στην έκθεσή του βλέπουμε πραγματικά που βρισκόμαστε. Έχω όμως και τρία σχόλια. Βάσει της εμπειρίας μας από τα τελευταία χρόνια, όσον ε, αφορά τα Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ή Κινητών Αξιών και Αγορών, έχουν γίνει διάφορες επαληθεύσεις και διαπιστώσαμε ότι η πίεση ήταν όλο και μεγαλύτερη πάνω στο προσωπικό. Και αυτό ε, προερχόταν η πίεση αυτή από τον νομοθέτη. Μα εμείς ε, ψηφίσαμε αυτό το δικαίωμα παρέμβασης. Δεν θα έπρεπε όμως να καταλήγει και σε εμπόδια, σε κάτι το οποίο να δυσκολεύει το έργο των αρχών αυτών. Η ΟΠΑ πιστεύω ότι έτσι καλλιώς πρέπει να είναι σε θέση να κάνει τη δουλειά της, κυρίως μάλιστα όταν πρόκειται για φακέλους, για τους οποίους εγώ μερικές φορές ήμουνα αξιολογητής. Μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι ξεπερνιέται το στάδιο της αρχής ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντέξεων. Ο πρόεδρος αντέδρασε, απέρριψε τις ε, προσφυγές ε, που έγιναν, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τελικά που είναι το πρόβλημα. Όσον ε, αφορά την ΕΣΜΑ, θα πρέπει εμείς ως νομοθέτες να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι νομοθετικές αρχές κατά προτεραιότητα και για τις τρεις αρχές βασικά. Για την ΕΣΜΑ θα πρέπει η λειτουργία του οργάνου να βελτιωθεί τα πρώτα χρόνια τα πράγματα είχαν τοποθετηθεί καλά. Σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι επανέρχονται δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Από την αρχή που δημιουργήθηκε υπήρξε μια εποπτική αρχή, εποπτική τραπεζική αρχή, η οποία εποπτεύεται ότι γίνεται στις τράπεζες. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για τα νομισματικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε. Τώρα όμως πρέπει να αναρωτηθούμε ποια θα πρέπει να είναι η μορφή αυτής της τεχνικής αρχής. Ουσιαστικά είναι τρεις που πρέπει να μας δίνουν συμβουλές που θα μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις εμείς και η Κομισιόν. Ρωτάω λοιπόν, από ποια στιγμή και μετά μπορούμε να προβλέψουμε να ενσωματωθεί η δομή αυτή με συνοχή στο όλο σύστημα, ώστε να λειτουργεί χωρίς ε, προβλήματα και χωρίς αντιφάσεις μεταξύ των αρχών. Φυσικά. Και πρέπει η αρχή που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο να μετεγκατασταθεί, εννοείται, εφόσον μιλάμε για Brexit. Υπήρξε όμως ένα συμβόλαιο ενοικίασης που υπογράφηκε και ισχύει μέχρι το 2026 και προβλέπονται κυρώσεις αν δεν τηρηθεί το συμβόλαιο αυτό και θα μας κοστίσει πολλά εκατομμύρια. Οπότε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε στενά. Το ελεγκτικό συνέδριο με τα στο αναφέρει. Δεν φτάνει. Υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να βελτιωθούν για να μπορούμε έγκαιρα να παρεμβαίνουμε. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή που το αναφέρει στην έκθεσή του. Δεν ε, βοήθησε το πνεύμα του ελεκτικού συνεδρίου, πάντως ανησυχούμε. Αυτά για την απαλλαγή για τις τρεις αυτές εκθέσεις. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογο. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Α, α ο εισηγητής, άντε, πω, πω, σε ξέχασα, συγγνώμη. Σύντομο όμως, έτσι. Η χρηματοδότηση και αρμοδιότητες είναι κυρίως τα θέματα. Και πώς θα μετεγκατασταθούν οι αρχές, ε, κάτι που δεν είχαμε προβλέψει. Σίγουρα θα έχουμε ενδιαφέρουσε ε, συναντήσεις. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Ωραία. Προθεσμία λοιπόν για την υποβολή τροπολογιών 17 Ιανουαρίου. 12 το μεσημέρι εν μέσω εκλογών. Τότε είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ο Σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ έχει όμως μια ερώτηση. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Πότε θα ανοίξει η διαδικασία για να μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Πότε μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Δεδομένου ότι ακριβώ έχουμε εκλογέ την επόμενη εβδομάδα, είναι λίγο περίεργο. Έχουμε μόνο τρει ώρε να το συζητήσουμε. Πότε, αύριο από αύριο μπορούμε να καταθέτουμε τροπολογίε. Τώρα. Τη Δευτέρα ταξιδεύουμε έτσι κι αλλιώ, ε, οπότε πήγε γιατί υπάρχει και εσωτερική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ωραία, θα ανοίξει το σύστημα ήδη αυτή τη βδομάδα, ναι. 6 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. 27 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Στην Επιτροπή Προπολογισμών ψηφίζουν 23 Μαρτίου, οπότε όλα θα πρέπει να, ε, να είναι έτοιμα, αλλιώς δεν θα παίξουμε κανένα ρόλο στην ψηφοφορία τους. Και Στη συνέχεια, τον Απρίλιο στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και φτάνουμε στο σημείο 9 που πρόκειται για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Επενδύσεων και Κεφαλαίων Κινδύνου. Η κυρία Πιέτικα σε πέντε λεπτά θα φτάσει από ό,τι μου λένε, οπότε τρία λεπτά διάλειμμα. Κανείς δεν είναι εδώ. Μικρό διάλειμμα λοιπόν.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 Yeah, Κυρίες και κύριοι, μόλις έμαθα ότι ο αντικαταστάτης της εισηγήτριας βρίσκεται εδώ στην αίθουσα, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε και λυπάμαι που διακόπτω τα πηγαδάκια σας. Συνεπώς, σημείο 9. Ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Απέτη Κάινεν πρώτα απ' όλα ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ και να παρουσιάσει η ίδια. Είχε προσωπικές υποθέσεις που την ανάγκασαν έκτακτες, που την ανάγκασαν να επιστρέψει στην Φιλανδία προτείνει τρεις αλλαγές η Κομισιόν στους κανονισμούς που καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κινδύνου και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Πρώτα απ' όλα, το εύρος των διαχειριστών για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δεύτερον, αυξάνεται και αριθμό των επιχειρήσεων όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις από αυτά και τρίτον η καταγραφή των ε, ταμείων γίνεται πολύ πιο εύκολα πια και πιο φθηνά. Η κυρία Πίτικάινεν στηρίζει τις προτινόμενες αυτές αλλαγές, αλλά θα ήθελα να δει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτά τα δύο ευρωπαϊκά πλαίσια. Πρέπει να τα δούμε γενικότερα στα πλαίσια της Ένωσης Κεφαλαίου Η μεγαλύτεροι αριθμοί στις τροπολογίες της έχουν να κάνουν με τα σημεία καταγραφής των ταμείων αυτών. Και θα ήθελε η ΕΣΜΑ να αναλάβει τις ευθύνες της επ' αυτού. Οι δύο κανονισμοί πάντως έχουν ενιαίους κανόνες για τις δύο κατηγορίες για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση ενισχύεται ακόμα περισσότερο εφόσον η ΕΣΜΑ έχει την ευθύνη της καταγραφής των ε, ταμείων αυτών. Έπειτα η έκθεση προτείνει σε αυτό το σημείο η ΕΣΜΑ να αναλάβει την καταγραφή. Πολλές χώρες μέλη βέβαια θα έχουν την, ε, το καθήκον της εποπτείας. Συζητήσαμε όλες και όδες με την κυρία με την συγγήτρια και όλοι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να υπάρξει αυτή η διεύρυνση και βέβαια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ απόψει σας. Τώρα για την πρόταση της Επιτροπής για την απαγόρευση των τελών που θα μπορούσαν να επιβάλλονται στα ταμεία αυτά από τις αρμόδιες αρχές των ε, χωρών ε, μελών, στηρίζουμε την απαγόρευση αυτή. Κύριε είναι στην έκθεσή της θέλει επίσης επιπλέον διευκρινήσεις ώστε τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας να ασχολούνται και με τις αγορές και την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένα τέτοιο ταμείο σε μια χώρα θα μπορεί και να εμπορεύεται και να διαχειρίζεται ταμείο σε άλλη χώρα μέλος. Οι διαχειριστές θέλουν να μπορούν να διαχειρίζονται ταμεία σε άλλες χώρες μέλη που θα εμπίπτουν βέβαια, θα συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς. Μιλάμε λοιπόν για ένα διαβατήριο κατά κάποιο τρόπο και για την ε, αγορά και για την διαχείριση. Είναι εξάλλου ένας από τους στόχους της ε, Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. είπαμε ότι θέλουμε η ΕΣΜΑ να καθορίζει, λέει η Επιτροπή, τα σωστά επίπεδα, ενώ η κυρία Πετικάνεν λέει να είναι αυτό μόνο για την περίπτωση κάτω από 250 εκατομμύρια. Για μεγαλύτερα ταμεία θα πρέπει να καθοριστούν και ήδη οι πόροι, ίδια ταμεία. Τέλος, δύο άλλες αλλαγές προτείνει η κυρία Πετικάινεν που όμως είναι μόνο για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Να υπάρξει χαμηλότερο όριο για τις ελάχιστες επενδύσεις στο Ιούσεφ, από 100.000 σε 50.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το όριο των 100.000 ευρώ ελάχιστο ποσό για να μπαίνει κανείς μέσα για μη επαγγελματίες επενδυτές μπορεί να ισχύσει για μικρότερα ταμεία. Το ΓΕΣΕΦ όμω, το Ταμείο Αυτό Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, είναι έτσι κι μικρό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να χαμηλωθεί το όριο, να μειωθεί, ώστε να ευνεθούν περισσότεροι ενδυνάμοι επενδυτές. Η πρόταση αυτή επίσης θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάποιες προτάσεις για προστασία. Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με το ενεργητικό και με τον ορισμό του θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε ποσοτικά το κέρδος αυτό. Αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Η συγκήτρια θέλει να ξέρει τις απόψεις των συναδέρφων για την έκθεσή της και να συζητηθούν παρετέρω οι ιδέες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Οι σκιώδεις μας τώρα. Αντρέα Κοτσολίνο πρώτα από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ, Αντρέα. E Ευχαριστώ τη συνάδελφο για τη συμβολή της και την προσπάθεια που έκανε να ληφθούν υπόψη οι ανταγωνιστικέ ανισότητε μεταξύ των χωρών και να αναθεωρηθεί η σχετική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική η αγορά. Έχουμε χρόνο να ε, καταρτήσουμε τη σωστή τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το θέμα. Τι εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Να θυμίσω αυτά που είχε και η κυρία Σεπτέμβριο για την ε, εκτίμηση μου προ το έργο τη Επιτροπή για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό σε γραφειοκρατικό επίπεδο για τι περιπτώσει ε, των ταμείων και των εταιριών που συζητάμε και για να υπάρξουν περισσότερε επενδύσει. Θα πρέπει να προσθεθούν κάποια στοιχεία που ε, να αποτελέσουν και αντικείμενο τοπολογιών φαντάζομαι, για να βελτιωθεί το κείμενο. Κυρίως η πρόταση τη Επιτροπή ώστε η ΕΣΜΑ να αναλάβει τη μέθοδο απολογισμού για το επίπεδο των κεφαλαίων που θα πρέπει να προβλέπονται. Θα πρέπει εδώ να ε, περιληφθεί αυτό στον ίδιο τον κανονισμό χωρίς να περιμένουμε η ΕΣΜΑ και η ΕΜΠΑ να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να υπάρχει ήδη νομική βεβαιότητα και δικαιοσύνη χωρίς να περιμένουμε ακόμη ένα χρόνο. Επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει να μην επιβάλλονται προμήθειες από την πλευρά των ε, αρχών ε, επίβλεψης που βρίσκονται στη θέση της υποδοχής. Αυτό ε, εξαρτάται από την ανάπτυξη της δράσης και της γεωγραφικής κάλυψης των αρχών. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε όταν θα υπάρξουν τέλη και να το εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές προβλέποντας ένα κατάλληλο σύστημα εφόσον χρειαστεί. Ε, επίσης για την αναλογικότητα, οι μικροί επενδυτές θα πρέπει να έχουν ακόμη πιο απλοποιημένη πρόσβαση. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σύστημα κάπως πιο light, πιο ελαφρύ. Σε αυτό το σκοπό, προς αυτή την κατεύθυνση, θα εργαστούμε το επόμενο 15 ώστε να καταλήξουμε σε μια εκδοχή του κειμένου, με την οποία να μπορεί να συμφωνήσει και η συγκέντρια και εμείς. Ευχαριστούμε για τους φιλελευθέρους. Για τους φιλελευθέρους. Η κόρα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω από τον κύριο Μπάλης να μεταφέρει τα συγχαρητήριά μου προς την εισηγήτρια για όλες τις προσπάθειες της σύνταξη αυτής της έκθεσης. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να προβλεφθούν πηγές χρηματοδότησης ποικίλε από τις ε, εταιρείες της νεόφυτες μέχρι τις μογκολιθικές. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η χρηματοδότηση θα υπάρχει σε όλες τις φάσεις, πράγμα που γίνεται θα πρέπει να γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως γίνεται και στην Αμερική. Θα πρέπει επίσης ε, τα δύο αυτά σήματα να είναι ελκυστικά ώστε να προσελκύουν χρηματοδοτήσεις ε, και να λειτουργούν καλά σε όλα τα στο Γιούσεφ. Ακόμη δεν ικανοποιήθηκε η υλοποίηση και αυτό το έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως με, την, ε, με τον σωστό καθορισμό του χαρτοφυλακίου των εταιριών σε στιγμή της ίδρυσής τους, κάτι που θα καθορίσει τα πράγματα και στο μέλλον. Επίσης, να καταργηθούν τα τέλη του κράτους υποδοχής. Σωστά το λέει αυτό η συγκήτρια και οι χρηματοδοτήσει να συνδυαστούν και με αυτό. Ε, η χρηματοδότηση σε συνάρτηση με το σήμα USEF είναι ένα σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι ακόμη μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν οι μη επαγγελματίες ε, επενδυτές μπορεί να επιλεγούν και για τις περιπτώσεις Γιουβέκα. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε αν θα περάσουμε σε άλλο ποσό από τα 500 από τα 100.000 και όλα αυτά ανυπομονώ να τα συζητήσω με την ομάδα των συγκητών ώστε τα δύο αυτά σήματα, ε, οι δύο αυτές μάρκες να ε, επιτρέψουν να τονωθούν οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά συνάδουν απολύτως και με το Μύθιξ. Πολύ ωραίο το τελευταίο που είπατε. Σας άκουγα. Τι λέτε. Για την ΚΟΕ. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, θεωρώ το συγκεκριμένο φάκελο πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί εντάσσεται σε μια συζήτηση που αφορά στην ενίσχυση πολιτικών ανάπτυξης στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ενίσχυση επιχειρηματικών projects τα οποία έχουν ε, κοινωνικό χαρακτήρα και προφίλ. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ήδη η έκθεση που αξιολογεί και τις επιπτώσεις από την μέχρι τώρα λειτουργία των δύο ταμείων, το περίφημο impact assessment, θέτει ψηλά τον πύχη έπειτα και από την αποδεδειγμένη με αριθμούς αποτυχία που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ε, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε από την Κομισιόν. Η εισηγήτρια, η κυρία Πετικάινεν, έχει κάνει αρκετή δουλειά μέσω των τροπολογιών που έχει καταθέσει και θα ήθελα και εγώ να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Ε, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα μέσα από αυτό το report να επιδιώξουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχήματα όπως ορίζονται μέσα από το eu και το EU-VECA. Ε, η οπτική με την οποία προσεγγίζω το θέμα ε, υπαγορεύει την ανάγκη μιας στροφής των ταμείων σε ένα μεγαλύτερο και πιο ευρύ φάσμα επενδυτών, ε, αλλά κυρίως μικροεπενδυτών, οι οποίοι είναι και αυτοί που ενδιαφέρονται να στηρίξουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίοι αυτή την περίοδο δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια ταμεία. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, το όριο πρόσβασης στα ταμεία Ιουσέφ ε, να κατέβει από το όριο των 100.000 ε, ευρώ και να κινηθεί προς την κατεύθυνση των 50.000 ευρώ. Αυτή είναι η δική μας θέση, αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε στην ε, μεταξύ των Σάντο Ραπορτέρς για να βρούμε την αναγκαία συνένεση και ισορροπία. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι και τα δύο ταμεία θα λειτουργούν με έναν τρόπο ε, πιο συνεκτικό, πιο διαφανή και γεωγραφικά πιο ισορροπημένο. Και θα πρέπει να δούμε και διαφοροποιημένα κριτήρια τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να ενισχύσουν και να ενσωματώσουν και μια εναλλακτική ε, λογική χρηματοδότηση σε projects κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικών επιχειρήσεων, να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και να ενισχύσουμε επενδυτές σε αυτόν τον ενδιαφέροντα και γεμάτο ε, ρίσκα και δύσκολο επιχειρηματικά τομέα. Από την άλλη πλευρά το EU10 θα πρέπει να γίνει πιο λειτουργικό για κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες. Θεωρώ για παράδειγμα ότι 499 εργαζόμενοι ή το όριο των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε assets είναι όρια απαγορευτικά για χώρες όπως η χώρα μου η Ελλάδα που έχει μεγάλη ανάγκη ειδικά αυτή την περίοδο για ενίσχυση ε, επενδύσεων. Όπως επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά τέτοιων projects και σε κλάδους και γεωγραφικά για να αποφύγουμε μια ακόμη φορά να γίνουμε μάρτυρες μιας κατάστασης όπου η πλειοψηφία αυτών των κεφαλαίων πηγαίνουν ε, σε αυτούς που τα έχουν και λιγότερη ανάγκη, στα χέρια λίγων managers από πλούσιες χώρες για να χρηματοδοτούν α, φαραωνικά καμιά φορά projects που δεν έχουν και ιδιαίτερη χρησιμότητα ή προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ενδιαφέρον για την κυρία Πετικάινεν για να συζητήσουμε και μεταξύ μας οι Σάντο Ραπορτές με την εισηγήτρια για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κανέναν από τους πρασίνους. Ας μιλήσει ο, ο, Φιλίπ. Νομίζω μάλιστα ότι είμαι και σκιώδης συγητής των πρασίνων για το θέμα αυτό. Σύμφωνα πάντως με όσα έχει ο πρόεδρος μπροστά του, δεν υπάρχει κανένας από τους πράσινους. Πρόεδρε, ε, κινούμε διακριτικά γι' αυτό, ώστε να, να είμαι κάτω από τα ραντάρ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Πιετικάινεν. Πώς είπατε? Ω, είμαι διαφανής, ναι, ναι. Συγχαρητήρια και στον Μπουρκχαρτ για την έκθεση για να υπάρχει το password και για το marketing και για το management συμφωνούμε και με την υποστήριξη της ε, εισηγήτριας για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση των ε, ταμείων που χρησιμοποιούν τις ε, ετικέτες UVSA και USEF. Να μπουν και κάποιες διαφυλάξεις μέσα με τη χρήση των σημάτων UVSA και USF να υπάρξει κάποιο ξεκαθάρισμα, να έχουν δηλαδή πραγματική ουσία. και για τις απαιτήσει για τα ταμεία, ώστε να διατηρηθεί μια αναλογικότητα ανάμεσα ε, σε ταμεία με κάτω από 250 εκατομμύρια και πάνω από αυτά και τις σχετικές απαιτήσει Ήδη το waiver έχει συζητηθεί στον πρώτο γύρο της συζήτησης USA και USF. Ήταν το κατόφλιο των επενδύσεων στα ταμεία αυτά και είχαμε πει καταρχήν 100.000 γιατί θέλαμε οι μικροί επενδυτές να αποφευθεί να μπουν σε υπερβολικά επικίνδυνα επενδυτικά ταμεία. Και είπαμε, αν είσαι retail investor, σωστό είναι να πάτε σε ένα να πάτε σε ένα τέτοιο ταμείο. Εάν, τότε όμως, υποφελείστε και από, τη, από τα προγράμματα προστασίας των επενδυτών των ταμείων usage ως ΕΚΑ. Εμένουμε στην θέση μας αυτή. Δεν θα πρέπει να μειωθεί το κατόφλι της εισόδου. Τώρα έχω και τρία πρόσθετα θέματα. Πρώτο, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επεκταθεί το φάσμα των επενδύσεων των ε, ταμείων. Σημειώνουμε την, την ε, ε, πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επενδύσεις εταιρείε μέχρι 499 εργαζομένους και το όριο των 50 εκατομμύριων που εξακολουθεί να είναι σημαντικό για μας. Σε ό,τι αφορά τα τέλη, υποστηρίζουμε την πρόθεση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή ε, τελών. Θεωρούμε ταυτόχρονα ότι οι ειδικοί κανόνες μπορούν να επιβάλλονται στον κανονισμό αυτό για να διέπουν τα τέλη τα οποία επιβάλλουν οι ε, μάνατζερ αυτού, οι διαχειριστές αυτών των ταμείων. Τέλος, τροπολογίες για να περιληφθούν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα μετρούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών. Και κάποια κριτήρια ή μπορούν πάντως να περιληφθούν και στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κεφάλαιου. Αυτά είναι οι τροπολογίες που προτιθέμεθα να καταθέσουμε και θα συνεργαστώ βεβαίως με τη ΣΥΡΠΑ. Thank you very much. I don't see any... Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κανέναν από την EFTD, ENF και πάλι δεν έχει οριστεί κάποιος. Κάτσε the τώρα. Η κυρία Τζίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ. Η πρόταση αυτή είναι σημαντική στα πλαίσια τη Νομισματική Ένωση. Διότι αν διηγείται τι γίνεται σε σύγκριση με τι ΗΠΑ και τι κεφαλαιοχικέ μα ενώσει, είμαστε στο 1 πέμπτο από τη δύναμη των ΗΠΑ αλλά έχει σχέση και με τη συζήτηση για τον προπολογισμό μα γιατί είναι το 6% του συνολικού κεφαλαι... της συνολικής κεφαλικής κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό. Άρα είναι σημαντικό πώς θα τονώσουμε την όλη δραστηριότητα. Και να βρούμε μια λύση εύχριστη, γιατί το θέμα είναι ότι η τωρινή πρόταση δεν εξετάζει το ζήτημα των τρίτων χωρών. Και αυτός θα ήταν ένας τρόπος να προτείνουμε κάτι παραπάνω. Η δεύτερη μου παρατηρήση έχει να κάνει με το ότι δεν είμαι βεβαία. Για το πώς όλο αυτό θα διοργανωθεί. Εδώ οι διαχειριστές είναι θέμα ότι ε, ρόλο θα αναλάβουν, το λέει και η αρχική πρόταση του κανονισμού και για να απαντήσω και στους συντονιστές δεν είμαι βέβαια ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ΕΣΜΑ. Και απλώς να μας αποσχολήσει η φάση της ε, καταχώρησης, της καταγραφής. Τη εισαγωγή, μάλλον, ε, πρέπει να δούμε και τη φορολογία. Διότι αυτό παρεμποδίζει μεγάλο μέρος τη ανάπτυξη σε σχέση με τα κεφάλαια κινδύνου. Δεν είναι η στιγμή τη εισαγωγή, λοιπόν, είναι διαφορετική η φορολόγηση. Αυτό πρέπει να δούμε. Για να μην υπάρχει κατακαιρματισμό. Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Very much. The next one on my list is... Η κυρία Παούνοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στηρίζω πολύ την υπόθεση αυτή. Έχω δουλέψει και εγώ πάνω σε αυτό για αρκετό καιρό και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τόσο πολύ την ανάπτυξη στην Ευρώπη που πρέπει να ψάξουμε να βρούμε οποιοδήποτε τρόπο για να τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για τις ε, κοινωνίες μας και για τις επιχειρήσεις μας να ανθίσουν. Με αυτόν τον κανονισμό αυτό που κυρίως μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τις δυνατότητες, να πάρουμε τα εμπόδια που υπάρχουν προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει η άνθηση αυτή. Είναι πράγματα που τα συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Πρέπει να γίνουν πιο αποφασιστικές δράσεις και όσο γίνεται πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο πάω σε συναντήσεις με επιχειρηματίες και ακούω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα όπως θα έπρεπε. Αν λοιπόν μπορέσουμε να τηρήσουμε ακόμα καλύτερα τις υποσχέσεις μας, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα θα βρεθεί συνένεση εδώ στο σώμα για να γίνει αυτό. Στηρίζω το κείμενο που διαγράφει τα τέλη που πρέπει να πληρώνουν στις χώρες υποδοχής ε, τα ταμεία αυτά. Θέλω να αναφέρω και κάποια νούμερα, γιατί εκπλήσει το γεγονός ότι κάτω από 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι τα κεφάλαια ψηλού κινδύνου, ενώ στι Ηνωμένε είναι παραπάνω. Οπότε προκειμένου το χάσμα να μειωθεί και κυρίως για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τον κλάδο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εξετάζουμε τάζουμε επίμαχα μέτρα όπως είναι οι ελάχιστες επενδύσεις ε, που χρειάζονται κτλ. Γι' αυτό και χαίρομαι με την πρόταση της εισηγήτριας που θέλει να μειώσει το ελάχιστο ε, ποσό για να μπει κανεί σε τέτοιο ταμείο. Ελπίζω να πετύχουμε ένα κείμενο το οποίο να ανταποκρίνεται θετικά απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα και επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Η Θερμάνος Μπέρε είναι η τελευταία ομιλήτρια πριν ξαναδώσουμε το λόγο ε, στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος ε, Φατζουλίνο. όλες τις παρατηρήσεις, άκουσα και την Ινα και έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, όταν το καθεστώ αυτό δημιουργήθηκε, ήταν πριν να έχουμε την έννοια της Ένωσης Κεφαλαίου Γνωρίζαμε τον κίνδυνο και τους περιορισμούς. Ο περιορισμός είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη κινητοποίηση των κεφαλαίων κινδύνου υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν υπήρχε ενιαία κεφαλαία αγορά και αυτό ήταν ένα μειονέκτημα για την καινοτομία κλπ. Απ' την άλλη όμως, δημιουργώντας τέτοια καθεστώτα, γνωρίζουμε ότι δημιουργούμε κάποιους θύλακες με κίνδυνο παράκαμψης κάποιων αρχών και κάποιων επιπτώσεων παρενεργειών που μπορεί να είναι βλαβερές. Γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες και συμφωνώ σε πολλά με την εισηγήτρια όσον αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση είμαι πολύ επιφυλεκτική για να μειωθεί το αναγκαίο κεφάλαιο για τα ταμεία αυτά. Γιατί αλλιώς στρεβλώνεται η κατάσταση, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση με αυτό που συνολικότερα θέλουμε να κάνουμε, που είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια και άρα δεν αναλαμβάνουμε υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο. Το να αναθέσουμε στην ΕΣΜΑ την ομοθεσία για το όριο του κεφαλαίου δεν με βρίσκει σύμφωνη. Σέβομαι πάρα πολύ την ΕΣΜΑ και πιστεύω ότι είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη για να ε, βοηθάει και να συζητάει με όλους τους παίκτες της αγοράς. Αλλά όταν δεν καταφέρνει ο νομοθέτης να το κάνει, κανονικά ό,τι μπορεί να γίνει νομοθετικά πρέπει να γίνεται νομοθετικά. Θέλω λοιπόν κατανομή το ρόλο, δηλαδή ο νομοθέτης να αναλάβει τις ευθύνες του, να καθορίσει ποια είναι τα απαιτούμενα κεφάλαια σε αναλογικό επίπεδο και στη συνέχεια η ΕΣΜΑ να αναλάβει τα υπόλοιπα, την εφαρμογή δηλαδή και την εποπτεία. Για το πεδίο της νομοθεσίας, όπως και η συγγήτρια, έτσι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αναθεώρηση αυτή για να ενισχύσουμε την προστασία των επενδυτών, αλλά και για να φροντίσουμε το εργαλείο αυτό να εξυπηρετήσει τη χρηματοδότηση των στρατηγικών μας στόχων ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μακροπρόθεσμες επενδύσεις και υπέρ της οικολογίας. γιατί δεν πρέπει να γνωρίσουμε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν πρέπει να υποφεληθούμε από την νομοθεσία αυτή και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. να ευχαριστούμε. Ο συγκεκριτής μας τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες και όλους τους εισηγητές και άλλους που μίλησαν για τις παρατηρήσεις τους έθεσαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Συνολικά νομίζω θα μπορέσουμε τελικά να συγκλίνουμε. Βέβαια κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν στις λεπτομέρειες, ιδίως ό,τι αφορά τον ρόλο του ΕΣΜΑ. Τα ακούσαμε αυτά ιδίως από τις κυρίες εδώ ε, προς τα δεξιά μου, τις κυρίες Περόνς και Νίνα. Αυτό που έχει σημασία εν τέλει είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και μια ρύθμιση η οποία στην πράξη να υποστηρίξει τον κλάδο στο σύνολό του και να προσφέρει κίνητρα για ανάπτυξη ακόμα περισσότερα από ό,τι έως τώρα. Από την άλλη πλευρά, και εδώ θα συμφωνήσω με την Περβάνς Μπερές, ότι είναι σημαντικό στο μέλλον να είναι εξασφαλισμένη η στερεότητα των ταμείων. Αυτό είναι must. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει η ορθή κατανομή των ρόλων. Νομίζω ότι είναι θετική η έκθεση της ΣΥΡΠΑ Πιετικά είναι και τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι στο όνομα της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. 24 Ιανουαρίου προθεσμία καταθέσεως των τροπολογιών. Θα έχουμε χρόνο για την ε, διαδικασία απαλλαγή. Θα συναντηθούμε ξανά στις 26-27 Φεβρουαρίου για το θέμα αυτό. Η δε ψηφοφορία ελπίζω να μπορέσουν να συμφωνήσουν και οι σκιώδεις ιδέες. Θα περιμένουμε τις τροπολογίες βέβαια. Προβλέπεται τέλη Μαρτίου. 22-23. Ευχαριστώ λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε στο υπαριθμό 10 θα δώσω τον, ε, την ε, διεύθυνση στον Γαβριήλ Μάτο. Okay, thank you. Sir. Hello to everybody. Um, all the best for... Καλημέρα σε όλους. Καλή σας χρονιά. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Έχουμε 10 λεπτά, έτσι. Έρχονται οι συγκητές. Yok, tam ben Yeah. Okay, we can restart as 11.15 the time. Είμαστε ήδη 11 και 4. Θα συνεχίσω ισπανικά, λέει ο πρόεδρος. Σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση 2016. 437 τροπολογίες. Η συγγήτρια έχει ετοιμάσει πολλές συμβαστικές τροπολογίες που νομίζω ότι καλύπτουν περίπου όλες τις τροπολογίες. Οι σκιώδες ηγητές ε, συναντήθηκαν και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Χούμπνερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Λέει κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αρχίσω με μια διόρθωση. Κάθε άλλο παρά όλες τις τροπολογίες έχουμε καλύψει με τις συμβαστικές μας. 29 έχω ήδη, ίσως 31 ήδη να είναι οι συμβαστικές, τις οποίες έχουμε καταλήξει. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και πολλές ε, τροπολογίες. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι αδύνατον ε, να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες για όλες. Το να κάνει κανείς συμβαστικές σε αυτό εδώ το θέμα είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε κοινέ πολιτικές γραμμές ε, στις ε, τροπολογίες. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι απόψει και μέσα στις ίδιε τι πολιτικές ομάδες. Οπότε η προσπάθειά μας με τις συμβαστικές ήταν ακριβώς αυτό, να υπάρχει μια συνοχή, δηλαδή να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν και να καταλήξουμε έτσι σε μια συμβαστική πρόταση που να έχει όμως συνοχή. Συζητάμε σήμερα όπου ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά με τους σκιώδεις εισηγητές όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνάντηση επίσης και θα καταφέρουμε, πιστεύω, να διευκρινίσουμε και διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ακόμα στις συμβαστικές και στην επόμενη συνάντησή μας που θα είναι στο Στρασβούργο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 25 του μηνός. Θα σας αναφέρω κάποια ζητήματα πάνω στο οποίο έχουμε πετύχει συμβαστικές προτάσεις. Σημαντικά αλλά και δύσκολα συγχρόνως. Είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο για συμβαστική τροπολογία είναι η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το πώς ε, μπορούμε να επωφεληθούμε από την ένωση αυτή και πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη διάγνωση. Ξέρουμε ότι όλους μας απασχολεί αυτό. Το θέμα της αφαιρεγγιότητας, είναι ένα σωρό θέματα αυτά ε, γύρω από τα οποία μπορούμε να έχουμε μια κοινή γραμμή, εξού και συμβαστική. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διαφορές απόψεων, κυρίως για το χρονοδιάγραμμα. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο πήγε. Άλλοι πάλι λένε χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε λύσεις. για τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε καταλήγουμε σε κάποια συμφωνία. Μιλάμε και για την συμμετοχή του ευρωπαϊκού επίπεδου. Στα πλαίσια όμως των εθνικών νομοθεσιών, γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την εθνική νομοθεσία, εδώ νομίζω ότι ακόμα και τις αρχικές συμβαστικές τις κάναμε πιο ισχυρές αναφέροντας τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαστε κοντά, λοιπόν, σε συμβαστικές προτάσεις για αυτά τα θέματα. Το δεύτερο, ο δεύτερος τομέας, δεύτερη περιοχή όπου προσπαθούμε να πετύχουμε συμβαστική τροπολογία είναι το δημόσιο χρέος. Εδώ έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες για το δημόσιο χρέος των χωρών και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποια είναι η θέση των ομάδων. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώσαμε τις τροπολογίες που αναφέρουν τα ωφέλη, τους κινδύνους, ανάλογα βέβαια και με την εποπτική μεταχείριση. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου περιμένουμε ακόμα αποτελέσματα από το FSB που δουλεύει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς δεν θα καταλήξουμε σε μια οριστική θέση γι' αυτά. Χτενίζουμε τις συμβαστικές, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό. Συζητάμε επίσης τις διεθνείς ε, προδιαγραφές. Βασιλεία. Εδώ έχουμε το δίλημα κατά πόσο πρέπει να αναφέρουμε ισχυρά την ανάγκη να παραπέμψουμε πάντα στα διεθνή πρότυπα. Κατά πόσο πρέπει ή όχι, ή κατά πόσο μπορούμε να επιτρέψουμε την απομάκρυνση από τα διεθνή πρότυπα. Εδώ έχουμε συμφωνήσει, αν μη τι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να επηρεάζει το έργο που γίνεται για τα διεθνή πρότυπα. ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε και αν δεν μας ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα να μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτά. Μας ικανοποιεί αυτή η διατύπωση. Και επίσης είμαστε στην ίδια γραμμή και όσον αφορά τα διεθνή φόρα. Και εδώ χρησιμοποιούμε την πρόταση της Γκουλάρ. Θα τις προτείνουμε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί στη διατύπωση. Ελπίζω ότι θα το δεχθεί. Επίσης δεν έχουμε μεγάλες διαφορές για τις εθνικές επιλογές και τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και την ιεράρχησή τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Και υπάρχει και το πρόβλημα του too big to fail. Εδώ επαναλαμβάνουμε τη δυσαρέσκειά μας με την κατάσταση σήμερα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε όσο γίνεται πιο αντικειμενικά για να πετύχουμε πρόοδο. Αλλά βέβαια υπάρχει και ο περίφημος ελέφαντας ε, στο δωμάτιο που μπλοκάρει τα πράγματα. Φοβάμαι πάντως ότι εδώ ένα σεβασμός θα είναι εύθραυστος. Θα δούμε. Προσπαθούμε πάντως και συμφωνούμε όλοι σε αυτό ότι για το MIFID δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε, δεν πρέπει να το ξανανοίξουμε. Οι πράσινοι και θα ετοιμάσουν κάποια συμβατική πρόταση για μια νέα παράγραφο για το Brexit. Θα υπάρχει λοιπόν άλλη μια συμβαστική πρόταση που νομίζω ότι εύκολα θα δεχτούμε. Περιμένω και μια συμβαστική πρόταση από τους πράσινους και τους σοσιαλιστές για μια νέα παράγραφο όσον αφορά τις μακροεποπτικές πολιτικές. Περιμένουμε τις προτάσεις που μας υποσχέθηκαν. Νομίζω λοιπόν ότι καλά πάμε για να έχουμε συμβαστικές για το κείμενο, αλλά σίγουρα θα παραμείνουν και πολλές τροπολογίες που θα πρέπει να ψηφιστούν επιπλέον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, η πρώτα, τέσσερα λεπτά ο καθένας από τους σοσιαλιστές, Ντελβό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Τανούτα Χιούμπνερ διότι πραγματικά έδειξε πνεύμα ε, διάθεσης μάλλον διάθεση να εξεύρουμε συμβαστικές τοπολογίες και να συμβαστούμε. και στις συναντήσεις σχεδόν που είχαμε, οι συζητήσεις μας κάλυψαν όλες τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που ενδεχομένω να είχαμε. Μαζί με τους πρασινούς θα φροντίσουμε να ετοιμάσουμε την τροπολογία, να συντάξουμε την τροπολογία για την μακροοικονομική, την μακροεποπτεία και ελπίζω να προλάβουμε να την αποστείλουμε σήμερα κιόλα. Είναι πολλές οι τροπολογίες και αν τη διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρέπει να επανέλθουμε στην ουσία του θέματος εάν θέλουμε η έκθεση να επιδιώκει το στόχο της. Δηλαδή να στελεί ένα μήνυμα και να επιδιώκει ακριβώς μια επισκόπηση του πώς έχει προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση. ώστε να συνδυαστούν τα διάφορα νομοθετήματα που εγκρίνουμε. Πρέπει να πούμε τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά ή τι λείπει. Από την πλευρά των θετικών σημείων λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όντω επιτέλους ε, έχουν εφαρμοστεί από όλες τις χώρες οι συστάσεις σε μια χώρα, ότι βελτιώνεται η υποπτία, ότι κοινέ ομάδε επίβλεψη φαίνεται να λειτουργούν σωστά, όμως προφανέστατα υπάρχει το too big to fail. Δεν έχει απεληθεί εκεί το θέμα και λείπει και ο τρίτος και λείπει και ένα δημοσιονομικό backstop, το οποίο να επιτρέψει την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση για τι μεγάλε ε, αρχέ και την διάγνωση τη υγεία τη Τραπεζική Ένωση. Πρέπει όμω να φροντίσουμε να καλυφθούν τα κενά και οι ανεπάρκειε. Και νομίζω ότι όποιοι μα ακούν μα εμπιστεύονται για να βρούμε λύσει σε όλα τα θέματα που ε, προκύπτουν και μέσα στις ε, προβλεπόμενες προθεσμίες. Κάποια πράγματα συζητιούνται σε άλλο επίπεδο. Ξέρουμε και την πρόταση της Επιτροπής για το ΕΔΙΣ. Έχουμε την ε, ολοκλήρωση της Βασιλείας 3. Όλα τα πακέτα θα συζητηθούν. Να, ε, επισημάνω λοιπόν, δεν θέλουμε η περάτωση αυτών των δημοτεύσεων και συζητήσεων να προδικάζεται, να προβλέπεται ήδη από τώρα στην έκθεση αυτή. Είναι θεμητό ο καθένα να προσπαθεί να ε, σημαδέψει την ε, δική του περιοχή και γι' αυτό οι βουλευτές και εξωταμικευμένα και σε εβδομάδα προτείνουν τις τροπολογίες τους. Όμως για να είμαστε συνεπείς πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς χωρίς να ε, προδικάζουμε το, πόρι, το την έκβαση των συζητήσεων που γίνονται αλλού. Βλέπω την ανυπομονησία σας κύριε Πρόεδρε και τον εκνευρισμό σας. Θα σταματήσω εδώ. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο χωρίς να επηρεάσουμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν αλλού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είχατε και άλλο χρόνο. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Τάρμπατη. Ο κύριος Λούνες είναι σκιώδης για το θέμα αυτό και μου ζήτησε να ε, στείλω τις, ε, τη συγγνώμη του που δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Θα διαβάσω εκ μέρους του. Ο κύριος Λούνες θέλει να ευχαριστήσει την συγκήτρια για την εξέταση των συμμεταστικών τροπολογιών, οι οποίες οδηγούν σε αρκετά καλά σημεία ισορροπίας. Κατά τη διάρκεια της ε, ανταλλαγής απόψεων στην ΕΚΟΝ, ο κύριος Λούνες ζήτησε την συγκήτρια να απομακρύνει τον ξεχωριστό κύκλο για τη δυνατότητα ε, του δημοσιονομικού backstop από το σχέδιο έκθεση. και να παραμείνει σε τρία κεφάλαια. Ένα για το καθένα από τους ε, πυλώνε της Τραπεζική Ένωση. Χαίρεται που δέχτηκε αυτήν την αλλαγή στη δομή του κειμένου η Άλλε τροπολογίε των συνδετικών και μεταρρυθμιστών έχουν να κάνουν ε, με την έκθεση των κρατών, το too big to fail, με την πλήρωση των σωστών προποθέσεων πριν την έναρξη οποιοδήποτε, οποιοδήποτε συστήματο προστασία των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε ότι πολλέ τροπολογίε για τα θέματα αυτά έχουν υποβληθεί από άλλα μέλη και χαιρόμαστε που η συγγετρία έλαβε υπόψη ε, τι απόψει διαφορετικών ομάδων ε, στι συμβαστικέ τη τροπολογίε. Ω προ τον τρίτο πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση, όπω αναμενόταν, πολλέ τροπολογίε έχουν αποβληθεί ταυτόχρονα και πάνε σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι δύσκολο να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα σε ένα περιορισμένο αριθμό παραγράφων και με ανυπομονησία θα περιμένουμε τις προτάσεις της εισηγήτριας. Υπό αυτό το πνεύμα, ο κύριος Λούνες θέλει να παραπέμψει στο ΕΔΙΦ τη σχετική πρόταση και το σχέδιο έκθεση για εκείνο το θέμα που θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για την εξέβρεση συμβαστικών τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την υποδομητική συζήτηση για του συμβασμού με του εισηγητέ, του υπόλοιπου κοιόδη και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα είναι σαφή, φιλόδοξη και ρεαλιστική. Thank you very much. Ευχαριστώ. Από του φιλελευθέρου δεν με κάνει εδώ. Γκουε. Ο κύριο Ματ Κάρθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά τη Για τι συμβαστικέ τροπολογίε Και τι πολύ καλέ συζητήσει που είχαμε. Δυστυχώ δεν πήγα στην τελευταία συνεδρία των σχεδόν, δεν μπορούσα. Είχα ελληνικέ υποχρεώσει να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσεις, λοιπόν. Τα συγκεκριμένα θα τα πω με email. Αργότερα. Να καλωσορίσω τη δουλειά που έχει καλυφθεί ήδη από τι συμβαστικέ τροπολογίε, προκειμένου να εντοπίσουμε αιτία και ενδεχόμενε λύσει σε κάποιε περιπτώσει των εξυπηρετούμενων θεών και δανείων. Επίση, είναι θετικό δείγμα να υπάρξει καλύτερη διευθέτηση τη λειτουργία του τραπεζικού τομέα και θα πρέπει και η εφαρμογή της νομοθεσίας να μην γίνεται μόνο βάση ελαχίστων προκτήπων για το ε, και αυτό να μην βαρύνει μόνο τους φορολογουμένους. Θα πρέπει ε, αυτά όσο το δυνατόν περισσότερο να απαιτηθούν στην τελική μορφή της έκθεσης. Θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε την ε, χρόνια έλλειψη κερδοφορίας στην πλευρά του τομέα στην Ελλάδα να δούμε πώς επηρεάσαν οι πολιτικές λιτότητες και πώς το επενδυτικό πρόγραμμα ε, επηρέασε όλες αυτές τις διαστάσεις. Το κρατικό χρέος έχει οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις τα να χαλαρώσουν τις, ε, ε, τους κανόνες εποπτείας. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε για την επικίνδυνο. Εδώ θα πρέπει όλα αυτά να απεχθούν στην τελική μορφή τη έκθεση. Το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένε δυνατότητε να παρακολουθήσει του επόπτε το έργο του. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, υψώσουμε από κοινό τη φωνή μα. Ελπίζω η πρωτοβουλία αυτή να επιτρέψει να βρούμε τις κατάλληλες εμπαστικές λύσεις. Ε, το πιο σημαντικό είναι να γνωρίσουμε την πραγματικότητα ότι οι τωρινές περιορισμένες προτάσεις έχουν να κάνουν ε, με μια χαλαρή για την Ανατολική Ένωση και με το του fail που δεν έχει επιληθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις δραστηριότητες των μεγαλύτερων τραπεζών. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά αποδράσει για να ε, ξεχωρίσουμε τι τράπεζε επενδυτικέ και εμπορικέ. Αυτή η διάκριση βασικά πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε σωστά. Και έτσι ίσω να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του fail. Δεν ήταν πρόταση της αριστεράς αυτή, είναι πρόταση από την έκθεση του 2012 της ομάδας ε, υψηλού επίπεδου των εμπνευμόνων. Έχει μπλοκαριστεί για την ώρα, αλλά καλά θα ήταν να καλέσουμε σε επίτευξη πρόοδου. Αυτέ ήταν οι βασικέ μου προτάσει και αναμένω τη συνεργασία μου με την ε, συγκεντρία και του υπόλοιπου και Και τώρα για του πρασίνου, ο κ. Ουρτάσουν. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Νομίζουμε πάντως ότι ορισμένες παράγραφοι της εκθέσεως πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, διότι ο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι πάρα πολύ περίπλοκος και πολλές ε, ε τράπεζες ακόμη δεν έχουν επαρκή κεφαλαιακή κάλυψη. Θα πρέπει να φροντίσουμε για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεχόμαστε ότι ορισμένες από τις ιδέες μας έχουν και το εκτιμούμε ότι έχουν περιληφθεί στο πρώτο σχέδιο της, ε, της ε, εισηγητρίας ιδίως για τη ρύθμιση του ταχαίως ε, αυξανόμενου τραπεζικού τομέα και επίσης κανόνες για την συνετή διαχείριση. Βλέπουμε επίσης και το πνεύμα προθυμίας μέσα στην ομάδα διαπραγμάτευσης για να βρεθούν κάποιες λύσεις, ιδίως για την πώληση σε μικρούς επενδυτές τραπεζικών προϊόντων, θέμα πολύ σημαντικό για χώρες όπως η Ιταλία σήμερα, και επίσης το πλαίσιο prudential. επίσης πολύ σημαντικό και αυτό. Εμείς θα έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα το διανύμουμε σήμερα και να δώσουμε τέλος έμφαση σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για την έξοδο της ε, Βρετανίας να μην υπάρξει ε, όρια ανταγωνισμού. Ε, υποστηρίζουμε και ορισμένε τροπολογίε, τι οποίε έχουν υποβάλει και συνάδελφοι άλλων πολιτικών ομάδων. Συμφωνούμε, για παράδειγμα, ότι χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση στις ε, τράπεζες για να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να τους επιτρέψουμε να πτωχεύσουν. Mm. Το ίδιο για την Resolution Authority και για το MRL. Ε, υποστηρίζουμε ακόμα την έκκληση της Σιλβί Γκουλάρ για την λογοδοσία διεθνών ε, αρχών όπως η Επιτροπή της Βασιλείας απέναντι στην ΕΚΟΝ. Τέλος, θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι θέλουμε να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας για το χαμήλωμα των κατοφλίων για την Capital Guidance. Η, τα σχέδια τροπολογιών επιτρέπουν την χρήση της Capital Guidance για να προχωρήσουμε, όμως φαίνεται πως οι εποπτικές αρχές βάζουν έναν ήπιο πυλώνα για την Capital Guidance. Στις 27 Δεκεμβρίου το πρακτορείο Reuters είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ένα καθυστερημένο χριστουγεννιάτικο δώρο στην Deutsche Bank κατεβάζοντας από τα 10,76 στα 9,51% <clears throat> το κατόφλιο γλιτώνοντάς τους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ μιλώ για την Deutsche Bank ε, υπάρχουν λοιπόν ορισμένα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και αναμένω τη συνεργασία με τους άλλους και όλους Ευχαριστώ. Άλλοι σκιώδεις δεν υπάρχουν. Συνεχίζουμε με το Catch Η κυρία Πάουνοβα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ την κυρία Χύπνερ για την καλή δουλειά που έκανε ως τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης που αποτελεί καλή βάση για το έργο μας σε αυτόν τον τομέα που είναι βέβαια ευαίσθητος και περιπλοκός. Όλοι γνωρίζετε ότι ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές παραμένουν για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ορισμένοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο από τις χώρες μέλη. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε να ενισχύσουμε την νομισματική ένωση που χρειάζεται για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί ενεργώς στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης συμμερίζομαι ορισμένες ανησυχίες συναδέλφων και ιδίω ό,τι αφορά τον συντονισμό μεταξύ SRB και άλλων αρχών μέσα στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής εποπτείας, μάλλον χρηματοπιστωτικής εποπτείας, συγγνώμη, ορισμένοι <clears throat> θεωρώ ότι επικρίνουν υπερβολικά, χωρίς όμως να δίνουν και ξεκάθαρες λύσεις. Θα πρέπει να δώσουμε πιο ξεκάθαρες λύσεις. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η απελευθέρωση κεφαλαίου για επενδύσεις φροντίζοντας να απολυθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με όρους αγοράς. Αυτή είναι μια ανησυχία που μοιραζόμαστε πολύ. Και θα πρέπει να περιληφθεί σε ένα ξεκάθαρο, ισχυρό κείμενο εκ μέρους μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλος κανείς. Α, εσείς θέλετε, ναι. Ευχαριστώ. Ναι, καθυστέρησα να σηκώσω το χέρι μου αρχικά δεν ήθελα να παρέμβω σε μια διαδικασία που τα πάει καλά και που είναι σε πολύ ικανά χέρια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που βεβαίω τα πάει πολύ καλά μαζί με τους κοιόδης εισηγητές. Είναι πάντοτε πρόθυμη να συνεργαστεί αλλά και με τους άλλους απλούς βουλευτές και πριν από την κατάθεση των τροπολογιών και τώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Μου άρεσαν και αυτά που είπε η κυρία Ντελβό σχετικά με το ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία της εκθέσεως όπου αν μπούμε στις λεπτομέρειες των υποθέσεων, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα, ταχύτητες, αιρεσιμότητα, είμαι βεβαία ότι δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Τα είπατε και σε αυτά. Ακούγοντας και τι είπε ο κύριος Λόνες, μου φαίνεται λέει τα ίδια πράγματα περίπου. Λέει δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι η Τραπεζική Ένωση δεν είναι έτοιμη. Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκοί πυλώνες, ο τρίτο, δεν είναι ευρωπαϊκός, χρειαζόμαστε όμω ένα τρίτο πυλώνα. Άρα συμφωνούμε ότι είναι επίγον να ευρεθεί αυτό ο τρίτο, χωρί να μπούμε σε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Ευχαριστώ και την συνάδελφο του SND των Σοσιαστών και Δημοκρατών που το είπε αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται ότι Αυτά θα πρέπει λίγο πολύ να λέμε όλοι με μια φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος που να θέλει να πιάσει το μάτι μου δεν υπάρχει. Η κυρία Χιούπνερ. Συμφωνώ με την Εστέρ που μίλησε μόλις τώρα και η οποία συνόψισε στην ουσία την προσέγγιση που πρέπει να κρατήσουμε και να μην ανοίξουμε ξανά ζητήματα τα οποία ήδη έχουν κρυθεί όπως ε, η ε, πτώχευση των τραπεζών βασισμένη στις ε, ε οδηγίες της Βασιλείας κλπ. Και ακόμη δεν έχουμε λόγους να κρίνουμε ή να κάνουμε συστάσεις. Ας μπήμπουμε λοιπόν σε αυτό. Συμφωνώ με την ανησυχία αυτή. Το άλλο που θα ήθελα να θέσω το συζητήσαμε στην πρώτη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και ήταν σαφές από αυτά που έλεγαν οι συνάδελφοί μου ότι υπάρχει μια τάση να χώσουμε στην έκθεση αυτά, αυτή όλα όσα έχουν σχέση με τον τομέα και όλα τα προβλήματα των τραπεζών και στην Ένωση και ανά τον κόσμο. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση να αποφύγουμε να κάνουμε ένα είδο χριστουγεννιάτικου δέντρου που καθένα κρεμάει το στολιδάκι του αυτή την έκθεση. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της έκθεσης. Ελπίζω ότι θα κατανοήσουν και οι πολιτικές ομάδες ότι πρόκειται για σημαντική πρόκληση για την οποία προσπαθούμε να σεβαστούμε. Ε, βέβαια, καταθέτουμε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά δεν μπορούν να χωρέσουν όλα. Ως τώρα, τα όσα έχω εντοπίσει ως θέματα που μπορούν να μπουν στις συμβαστικές τροπολογίες, θα τα διαβάσουν οι συναδελφοί μου, να προχωρήσουμε με τη γραπτή διαδικασία πριν από την επόμενη συνεδρίαση, να κάνουμε μια ρύθμιση των λεπτομεριών, των συμβαστικών τροπολογιών. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου να δραστηριοποιηθούν στο ενδιάμεσο διάστημα πριν από την επόμενη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 25 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες, που έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις, που έχουν σχολιάσει και τα σχόλια αυτά τα βρήκα πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ Δανούτα. 25 Ιανουαρίου ψήφος. Θα δούμε για την Ολομέλεια. Φεβρουάριο-Μάρτιο. Διάφορα. Τίποτε στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου. Θα μετακινηθούμε τώρα στην αίθουσα 3 σε 50, στον τρίτο όροφο, όπου θα συναντηθούμε με την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ ΛΥΜΠΕ.